possiamo iniziare il nostro lavoro. Naturalmente ricordo... Θα αρχίσουμε νομίζω. Λοιπόν, λοιπόν ανακοινώσει. Θα κινηματογραφηθεί η συνεδρίαση και θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο. Και έχω ένα αίτημα όπου θα πρέπει δυστυχώς να επιστρέψω σήμερα στην Ιταλία και κατόπιν τούτου ε, δεν θα μπορέσω να παρουσιάσω την εκθέση που είχε προβλεφθεί για αύριο. Ε, η συνάδελφος Ραντζέλα ανταυτού έχει μπλοκαριστεί από το χιόνι και δεν θα έρθει σήμερα, θα έρθει αύριο. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να το αντιστρέψουμε στην ημερήσια διάταξη να κάνουμε μία αλλαγή. Δηλαδή της ε, κυρίας Ραντζέ, το θέμα που είχε προβλεφτεί για σήμερα το βράδυ, το 5 και το 6, αυτά να πάνε για αύριο και ε, η δική μου η ε, έκθεση να ε, μεταφερθούν σήμερα το απόγευμα, ελπίζοντας ότι μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα, διότι πρέπει να πάω στις 6 στην Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε ε, την ε, συνεδρία των συντονιστών στις 5. Αύριο το πρωί ε, οι συνάδελφοι που προβλέπονται δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου η πρόταση είναι στις 10 να ξεκινήσουμε, αντί για τις 10 να ξεκινήσουμε στις 10 και μισή ε, με τις ψηφορίες. Ε, αν λοιπόν ε, συμφωνείτε, ας ακολουθήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Γνωρίζω ότι το, η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών έχει ορίσει αναπληρωτή και δεν ξέρω αν είναι εδώ. Α, δεν είναι εδώ. Κατόπιν τούτου α, ε, να του, μπορούμε να του, εγώ θα του μεταβάσω τους χαιρετισμούς μου ε, με γραπτό τρόπο. Περνάω τώρα στις ε, ανακοινώσεις. Πρόκειται για, την, ε, για τον προπολογισμό του 2012 και εκεί υπάρχει μια ειδική επιφύλαξη της δικής μας της Επιτροπής. Κατόπιν τούτου, μετά από αυτήν την ανακοίνωση, τη δική μου την ανακοίνωση που αφορά στην συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου. Ο συνάδελφος Αντάρκας, ο δικός μας ο εισηγητής για τον προπολογισμό, έρθει σε επαφή με τον Γενικό Διευθυντή που είναι αρμόδιος για την πολιτική επικοινωνία, τον κύριο Γκρέγκορι Πούλβερ και ε, είχε αναλάβει και η κυρία Γκουρμάη, αλλά δυστυχώ είχε άλλε λιμένε υποχρεώσει και δεν μπορούσε να είναι παρούσα. Ε, κατ' ουσίαν λοιπόν συνέβη το εξή ότι οι ε, πληροφορίες που δόθησαν από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έπεισαν το συνάδελφο Σαουντάργας να αποσύρει τη δική μας την ε, επιφύλαξη ε, κυρίως όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό χώρο και με τον τρόπο αυτό αποδεσμεύτηκε το κονδύλι που είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. Ανταυτού ο εκπρόσωπός μας ε, στην Επιτροπή όσον αφορά άλλα κονδύλια και αναφέρομαι στο ε, κεφάλαιο εκείνο που λέει επικοινωνία με την ε, εταιρική σχέση, στο πλαίσιο της εταιρική σχέση, εκεί ο συνάδελφος Αντάργα είπε ότι δεν υπάρχουν, δεν δόθηκαν αρκετές ε, διευκρινήσει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η γραμμή του προπολογισμού. Κατά τα άλλα, σας προτείνω να δεχτούμε αυτά που προτείνει ο συνάδελφος κύριος ε, Σαουντάργας, ο οποίος ε, θεωρεί ότι όσον αφορά αυτό το δεύτερο θέμα είναι απαραίτητο να ακούσουμε την Αντιπρόεδρο κυρία Ρέντινγκ σε μία από τις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις μας. Αν λοιπόν συμφωνείτε κι εσείς, ας ε, ζητήσουμε με τη μορφή επιστολής ε, αυτό που σας είπα στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών και στην Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ να έλθουν να μας επιστηθούν σε μία από τις ε, επόμενες συνεδριάσεις μας. Από ό,τι βλέπω συμφωνείτε, ώστε τούτου έτσι θα πράξουμε. Πάμε στο 2-2. θα θυμάστε ότι υπάρχει ήδη η έκθεση Ταρκόφσκι. Δηλαδή υπάρχει έκθεση εκείνη με την οποία καλούμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ε, επικαιροποιήσουν την έκθεση που αφορά τη διαδικασία της συναπόφασης. Και στο θέμα αυτό, σύμφωνα με την έκθεση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνθήκη της Λισαβόνας, να διευρυνθεί, να διαδοθεί περαιτέρω η διαδικασία της συναπόφασης και κατόπιν τούτου να αναθεωρηθούν και οι δηλώσεις ε, που γίνονται στο Συμβούλιο, γιατί ε, κατά την άποψή μας ε, δεν θα έπρεπε να έχουν οι δηλώσεις αυτές καμία νομική βάση. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι αυτό είναι περισσότερο θέμα του ίδιου του Συμβουλίου και υπογραμμίζει η Επιτροπή ότι ε, θα ήταν ε, άκομψο να ζητήσει κανείς ε, παρέμβαση, διαθεσμική παρέμβαση, να το ζητήσουμε εμείς αυτή την παρέμβαση. Και αν ο συνάλφος Ταρκόφσκι θέλει να προσθέσει κάτι, βεβαίως μπορεί να το κάνει, από ό,τι βλέπω όμως δεν θέλει να προσθέσει τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Και θα ήθελα τώρα να ανακοινώσω ότι έχουμε εδώ και αντιπροσωπεία από την γερουσία της ε, Ολλανδίας που ζήτησαν να επισκεφθούν ε, μάλλον την Επιτροπή μας ε, στις 5 Μαρτίου. Και αυτή η συνάντηση έχει πάρει και ένα συγκεκριμένο τίτλο που λέει «Ευρώπη, που κατευθύνεσαι, εκβομπάντης» η συνάντηση ε, θα πρέπει να γίνει από τις 12.30 μέχρι τις 2.30 ε, ε, εδώ ή μάλλον καλύτερα στο Στρασβούργο, στο εστιατόριο των βουλευτών. Τα επιχείρηματα με τα οποία ασχολούνται οι Ολλανδοί είναι αυτά που ασχολούμαστε και εμείς. Δηλαδή, λόγω της κρίσης, οι σχέσεις που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια η επιλογή της ε, κοινωτικής μεθόδου για τις διακυβερνητικές σχέσεις, η ε, σχέση, η νέα διακυβέρνηση και η νέα οικονομική και νομισματική διακυβέρνηση. Οι δυνατότητες επιλογής ε, για μια νέα συνθήκη, η δυνατότητα μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων, κατά πόσο αυτό είναι εκταίο, όχι, Όποιος λοιπόν επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτό το μίνι συμπόσιο, ε, παρακαλείται να ε, το πει μέχρι την 1η Μαρτίου. Μέχρι τώρα ε, θα έχουμε, όχι 12, 6 μέλη του Κοινοβουλίου. Εγώ είπα 12, αλλά έκανα λάθος. 6 θα είναι τα μέλη και η συνάντηση θα είναι εδώ στις Βρυξέλλες, όχι στο Στρασβούργο. Σας ζητώ συγγνώμη. Πολύ ωραία. Πάμε ε, λοιπόν στο ε, χρονοδιάγραμμα των συναντήσεών μας και προτείνω μία ε, αναβολή. Η δική μας συνεδρία του Ιουλίου μεταφέρεται στις 11 το απόγευμα και στις 12 Ιουλίου το πρωί. Αυτή η τροποποίηση ήδη αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα ε, το οποίο ήδη σας έχει διανεμηθεί. Και εάν συμφωνείτε, σας ε, παρακαλώ να εγκρίνετε τα πρακτικά της 15ης ε, Δεκεμβρίου, τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. Εάν δεν έχετε καμία αντίρρηση, τα πρακτικά αυτά θεωρούνται ότι, θεωρείτε ότι τα έχετε εγκρίνει. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο, το 4. Πρόκειται για την ερμηνεία των άρθρων 48 παράγραφος 2 και 50 και τροποποίηση των άρθρων 20 και 27 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ είμαι εκείνο που θα κάνω την έκθεση. Άρα συνεχίζω. Αυτή λοιπόν η ερμηνεία προέρχεται από ερμηνεία 57 του άρθρου 57 του κανονισμού που έχει σχέση με την περίπτωση εκείνη κατά την οποία μία απόφαση, μία έκθεση απορρίπτεται από την Ολομέλεια ή αποσύρεται πριν φτάσει στο τελικό στάδιο του ε, ψηφίσματος. Στην περίπτωση αυτή, αυτή επανέρχεται στην Επιτροπή. Το πρόβλημα είναι τι, τι γίνεται ε, στην περίπτωση κατά την οποία είναι αρμόδιες περισσότερες επιτροπές. Συνέβη κάτι τέτοιο, όπου είχαμε συνεργασία με την Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών και φαινόταν ότι δεν υπήρχαν μεγάλα προβλήματα, γιατί ε, στην περίπτωση κατά την οποία η επί της ουσίας αρμόδια Επιτροπή δεν συμπεριλαμβάνει στη διαδικασία την ε, επιτροπή με την οποία συνεργάζεται, αυτό με βάση το άρθρο 50 η αρμόδια επιτροπή έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει στην Ολομέλεια την έκθεση και στην περίπτωση στην οποία αναφέρομαι κρίθηκε ότι ε, είχαν ληφθεί όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που αποδείκνυαν τη συνεργασία των δύο επιτροπών. Όμως προέκυψε μία επιστολή και ένα αίτημα κυρίως ε, του Προέδρου της ε, Επιτροπής, της Προέδρου, της κυρίας Μπερές, η οποία ζήτησε από τον ε, Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων ε, να, να εκφράσουν και αυτή την άποψή τους. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ε, πρόκειται βέβαια για ε, γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας. Με βάση το άρθρο 48, όπως ξέρετε πολύ καλά, εκεί προβλέπεται ότι είναι δυνατόν να κατατίθενται τροπολογίες μόνο όμως από τον εισηγητή της, επί της ουσίας αρμόδιας επιτροπής. Άρα λοιπόν, τίθε το ερώτημα. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εισηγητής της ε, Επιτουσίας Αρμόδης Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη του τις ε, τροπολογίες ε, της συνεργαζόμενης, ας την πούμε έτσι, Επιτροπής με βάση το άρθρο 50, τότε τι συμβαίνει, τι πρέπει να γίνει και πάνω απ' όλα σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας όπου με βάση το άρθρο 48 προβλέπεται η διαδικασία των τροπολογιών, τότε ισχύει το ότι ο εισηγητής της ε, συνεργαζόμενης επιτροπής έχει τη δυνατότητα να καταθέσει στην Ολομέλεια τροπολογίες ή όχι. Ποιο άρθρο υπερισχύει, το 48 ή το 50. Εδώ μας έχουν ζητήσει μία διευκρίνηση. Και με βάση ε, την αρχή, την Ιταλική ε, νομοθεσία. Νομ, στην Ιταλία ισχύει ότι η ειδική διάταξη υπερισχύει ε, της γενικότερης ε, διάταξης. Άρα δηλαδή υπερισχύει το άρθρο 50. Πρέπει όμως να αποφεύγουμε τις ασάφειες. Άρα δηλαδή πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή, κάποια τροποποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θέμα γενικότερης φύσεως, ε, στην περίπτωση κατά την οποία ε, διαπιστώνεται στη συνεργασία δύο επιτροπών ότι δημιουργείται αντίθεση και δεν καθίσταται δυνατόν να επιληθεί η αντίφαση αυτή, η αντίθεση ε, στη διάσκεψη των προϊόντων θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν προτείνεται να υπάρχει μια ερμηνεία, όπως ακριβώς αναφέρεται και στην επικεφαλίδα των άρθρων 48 ε, και 50, να τροποποιηθούν τα άρθρα 20 και 27, έτσι ώστε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, εφόσον το ζητήσει η διάσκεψη των πρόεδρων, να μπορεί να παρεμβαίνει, να ακυρώνει αποφάσεις ε, μιας ε, επιτροπής ε, η οποία δεν σέβεται την όλη διαδικασία και δεν σέβεται τη συνεργαζόμενη επιτροπή. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Ε, σας το παρουσίασα ε, όπως το σκέφτομαι εγώ και αν κάποιος βέβαια επιθυμεί να λάβει το λόγο αλλά από ό,τι βλέπω... Α, μισό λεπτό, ο κύριος Γκουαλτιέρη θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω μόνο να σας πω ότι η ερμηνεία την οποία προτείνετε εσείς είναι σωστή. Δηλαδή πράγματι αυτή η ιδιαιτερότητα που προβλέπεται στο άρθρο 48 αυτό που λέει το άρθρο 48 δεν μιλάει μόνο για ένα εισηγητή, αλλά μιλάει για τον εισηγητή γενικότερα ε, που σε ορισμένε ε, περιπτώσεις αυτό σημαίνει εξειδικευμένο εισηγητή για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Άρα δηλαδή εγώ πιστεύω ότι αυτά που λέτε είναι σωστά. Τα συμμερίζομαι. Και όσον αφορά τώρα, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε εμβαθύνει στο να εξετάσουμε αυτές ε, τις ε, τροπολογίες. Αλλά έτσι με την πρώτη ματιά ε, θέλω να σας πω ότι όσον αφορά το άρθρο 20 διερωτώμε κατά πόσον είναι τόσο σημαντική η τροποποίηση όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Προέδρου. Κατά πόσον αυτό μπορεί να εκλειφθεί ως ένα νέο άρθρο. Δηλαδή να υπάρχει πιο επίσημη ερμηνεία με την έννοια ότι το άρθρο 20,3 αφορά στη δυνατότητα να μπορεί ο πρόεδρος ε, στην Ολομέλεια να λαμβάνει το λόγο. Εδώ όμως ε, μιλάμε για κάτι το διαφορετικό. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι πρόκειται για το 3α. Δεν θα το έβαζα εδώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μου επιτρέψετε λιγάκι να το ε, σκεφτώ αυτό το θέμα, να δω ποια είναι η βέλτιστη λύση για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα που, όπως είπα, κατά την άποψή μου, ε, είναι κάτι το σημαντικό το οποίο λέτε. Εγώ δεν είμαι αντίθετος. Ε, κάθε άλλο, ξεφεύγουμε από, από το απλό θέμα της ερμηνείας του 48 και 50 και εισάγουμε μία εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου για θέματα τα οποία είναι πέρα από το αντικείμενο της έκθεσης, από το ε, περιορισμένο αντικείμενο. Θέλω λοιπόν ε, να πω ότι πρέπει να το σκεφτούμε λιγάκι όλο το θέμα. Εν πάση περιπτώσει εδώ ε, πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή η οποία ξεφεύγει, πάει πολύ πιο πέρα από το συγκεκριμένο θέμα ε, που αφορά την, ε, τις τροπολογίες 3 ε, και 4. Δεν ξέρω, αν δεν υπάρχουν... Μισό λεπτό, κύριος Χέφνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι μπορώ να είμαι σύντομος. Κοιτάξτε, και εγώ συμφωνώ με την ερμηνεία που δίνεται στους κείμενους κανόνες και την ερμηνεία σας τη βρίσκω και σωστή και λογική. Όμως θα μου επιτρέψετε να είμαι λιγάκι επιφυλακτικός όσον αφορά την ε, επιθυμία αυτή που εκφράστηκε για αλλαγή της όλης διαδικασίας. Γιατί νομίζω ότι το όλο θέμα ξεφεύγει λιγάκι από αυτό το συγκεκριμένο που συζητάμε. Εντάξει, δεν θέλω να αποφασίσουμε σήμερα, αλλά θέλω και εγώ να εκφράσω τις επιφυλάξεις μου. Τις επιφυλάξεις μου όσον αφορά την διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό στο καταστατικό προβλέπεται ως ένα συμβουλευτικό όργανο το οποίο μπορεί να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ε, η διάσκεψη των Προέδρων. Ε, όμως ε, εδώ προβλέπεται να έχει πολύ εκτεταμένες αρμοδιότητες. Το σημαντικό θέμα ε, νομίζω ότι ξεφεύγει από την ερμηνεία που δίνουμε και κατόπιν θεωρώ ότι όλο το θέμα χρήζει και περαιτέρω συζήτησης. Πολύ ωραία. Εντάξει, θα το συζητήσουμε, λέει ο Πρόεδρο, Θέλω να σα υπενθυμίσω ότι ήδη είναι αρκετά εκτεταμένες ε, οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου. Το άρθρο 20 λέει ότι ο Πρόεδρος συντονίζει τις ε, εργασίες ε, του Κοινοβουλίου και έχει την απόλυτη αρμοδιότητα για να μπορεί να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία η τροπολογία την οποία προτείνω εγώ είναι μια διευκρίνηση και λέει για να μπορεί να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου ο Πρόεδρος μπορεί με τη στήριξη της διάσκεψης των Πρόεδρων Αυτή λοιπόν είναι η αλλαγή που περιλαμβάνεται στο άνθρωπο 27. Μπορεί να λάβει τα απαραίτητα και τα κατάλληλα μέτρα. Αυτό λοιπόν είναι ήδη μια αλλαγή που αφορά στη, στη διάσκεψη των Πρόεδρων. Να λάβει λοιπόν τα απαραίτητα μέτρα που θα οδηγήσουν ε, στην ε, ακύρωση ενδεχομένως μιας απόφασης η οποία έχει ήδη ληφθεί. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει μία διευκρίνηση. Η απόφαση βέβαια του Προέδρου είναι ε, καταληκτική. Νομίζω ότι με αυτές τις παρατηρήσεις μπορούμε να κλείσουμε την όλη συζήτηση. Το μόνο που απομένει ακόμα είναι να ορίσουμε το πότε μπορούμε και πρέπει να καταθέσουμε τις ε, τροπολογίες αυτές. Εγώ τα έλεγα στις 22 ε, Μαρτίου, είναι καταληκτική ημερομηνία, σε 11 ώρα το πρωί, μέχρι τις 11 το πρωί, έτσι ώστε ε, το όλο θέμα να συζητηθεί στις 26 Απριλίου. Και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα αυτήν την έκθεση μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή να την παρουσιάσουμε και στη διάσκεψη των Προέδρων στην ε, Ολομέλεια του Απριλίου. Ε, αν συμφωνείτε, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στο σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις... Ε, σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίε του Λότ Ιρλανδίας όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο κύριος Ράντζελ είναι ο εισηγητής, αλλά είπαμε ότι αυτό θα πάει για αύριο το πρωί, όχι τώρα. Και ε, όπως έχουμε ήδη συμφωνήσει, πάμε στο επόμενο θέμα. Στο 12 το προτάξαμε για σήμερα είναι η ερμηνεία του άρθρου 117 εγώ πάλι θα μιλήσω γιατί δεν θα είμαι εδώ αύριο το πρωί. Πρόκειται για την ερμηνεία του άρθρου 117, παράγραφος 3 του κανονισμού, εξέταση των γραπτών ερωτήσεων σε επιτροπή. Κοιτάξτε, αυτό ε, νομίζω είναι ένα απλό θέμα. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μας ζήτησε τη γνώμη μας. Έθιξε εκείνη αυτό το πρόβλημα, δηλαδή πώς πρέπει να εφαρμόσει το άρθρο 117 παράγραφος 3 του κανισμού. Και ε, στην περίπτωση κατά την οποία αυτός που κάνει μια ερώτηση και δεν παίρνει την απάντηση μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, μπορεί να ε, ζητήσει το θέμα αυτό να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της αρμόδιας επιτροπής αμέσως μετά την εκπνοή της ημερομηνία. Έτσι λοιπόν, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, τότε προβλέπεται ότι η Επιτροπή, η Αρμόδια Επιτροπή ε, δεσμεύεται να ε, συμπεριλάβει αυτό το θέμα ε, στο οποίο αναφέρθηκα, αλλά καταλαβαίνετε εδώ θα υπάρξει ε, ένας ε, μεγάλος φόρτος εργασίας. Κατόπιν τούτου, εδώ, κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι έτσι μια γενική αναφορά στην ευελιξία, αλλά να υπάρχει μια συγκεκριμένη διάταξη του κανονισμού μία διάταξη η οποία θα δίνει αρμοδιότητα στους προέδρους των επιτροπών να μπορούν εκείνοι να καθορίζουν ε, την ημερήσια διάταξη. Αυτό νομίζω ότι είναι η σωστή ερμηνεία. Δηλαδή, μία ερμηνεία σύμφωνα με την οποία η ημερήσια διάταξη να ορίζεται σύμφωνα ε, σε συνεργασία με τον πρόεδρο και τον υποβάλλοντα την ερώτηση. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σήμερα. Και η Ολομέλεια μπορεί να ε, αναβάλει ένα θέμα ή να τροποποιήσει μία ημερήσια διάταξη. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι μπορεί κανείς να δώσει την εξής απάντηση. Είτε θα τροποποιήσουμε το άρθρο 117, να δώσουμε δηλαδή την απάντηση που σας ανέφερα, ή και σε αυτή την περίπτωση να προβλεφθεί τροποποίηση του κανονισμού έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση. Και σε αυτή την τελευταία περίπτωση πρέπει να γράψουμε στον ε, κανονισμό ότι στην επόμενη συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής αμέσως ε, μετά την ε, εκπνοή της προθεσμίας ε, μέσα στην οποία έπρεπε να δοθεί η απάντηση από την Επιτροπή. Δεν νομίζω όμως ότι βέβαια είναι απαραίτητο να γραφτούν όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Αλλιώς αν δεν ε, γίνουν όλα αυτά δεκτά θα πρέπει ε, να ε, συνταχθεί έκθεση. Ο κύριος Ταρκόφσκι. I have a very, very strong opinion on it, but uh, I have an opinion, which... Θέλω να σας πω το εξή. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να εξηγούμε τα πάντα στον κανονισμό μας. Θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο ευέλικτοι. Παραλαμβάνω λοιπόν, γιατί δεν νομίζω ότι με ακούτε κύριε Πρόεδρε, Παραλαμβάνω ότι δεν θα πρέπει να εξηγούμε τα πάντα στο κανονισμό, αλλά να τα ερμηνεύουμε. Να βλέπουμε δηλαδή ε, τους κανόνες. Λέμε εδώ ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίζει. Νομίζω αυτή είναι η καλύτερη λύση και επειδή προέρχεται από την ΑΦΕΤ, δεν νομίζω ότι κανεί μπορεί να αφισβητήσει το προνόμιο του Έλμαρ, είτε το δικό σα και έτσι γίνονται τα πράγματα ευκολότερα. Έχουμε όμω και τη δεύτερη εναλλακτική που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει αποδοχή ρητό από το πρόεδρο. Αυτό δεν νομίζω ότι δίνει την ίδια Και αν, όπω η ΑΦΕΤ, κατακλείζεται κανεί από όλα αυτά τα θέματα, τότε ο πρόεδρος Μπαίνει στον προβολέα, στο φώτο της δημοσιότητας, αν θέλετε, γιατί πρέπει, ε, άμα πει όχι, αυτό φαίνεται ότι το έχει κάνει αυτός, παίρνει όλη την ε, προβολή. Νομίζω λοιπόν ότι η πρώτη επιλογή, με βάση όλα αυτά που σας είπα, είναι καλύτερη από τη δεύτερη, για να μην έχουν και αλλαγή των κανόνων. Αυτή είναι η άποψή μου. Φαντάζομαι ότι είστε σε επαφή με τους ε, προέδρου των Επιτροπών, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή του, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ίδια με τη δική μου. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς, ε, επειδή άλλαξε η μερίσια διάταξη, η σκιώδη εισηγήτρια της ομάδας μας για αυτό το θέμα δεν είναι εδώ και δεν είχαμε και την ε, δυνατότητα να συζητήσουμε ε, για το θέμα αυτό γιατί θα έρθει αύριο. Γι' αυτό λοιπόν ε, εγώ ε, λαμβάνω το λόγο ε, επιθυμώντας όμως να έχω τη δυνατότητα να το συζητήσω το θέμα αργότερα με την ίδια την αρμόδια. Απλά θα πω έτσι την γνώμη μου με την πρώτη ματιά το άρθρο 193 υπερισχύει το 117. 193 υπερισχύει 117. Διότι όταν πρόκειται για μια επιτροπή η οποία έχει οριστεί από την πρόεδρο, αυτό το άρθρο το 117 με απόλυτη σαφήνεια δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του Κοινοβουλίου να υποβάλουν τις ε, ερωτήσεις τους ε, ερωτήσεις βέβαια για τις οποίες ε, δεν έχουν πάρει απάντηση, τις ερωτήσεις αυτές να τις εντάσσουν στην ημερήσια διάταξη μιας επιτροπής. Ε, εάν όμως αυτό γίνεται όπως ακριβώς, στην, ή μάλλον εμπίπτει στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής, τότε θεωρώ ότι αυτό δεν είναι σωστό και θα πρέπει πράγματι να αλλάξουμε τον κανονισμό. Δηλαδή να διευκρινίσουμε ότι το δικαίωμα αυτό εδώ θα έπρεπε να τροποποιήσουμε το άρθρο 117, δηλαδή να περιορίσουμε το δικαίωμα αυτό που έχουν ε, σήμερα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ε, με την έννοια ότι εδώ αναφέρεται όχι ζητούν να γραφτεί στη Μεσή Διάταξη, γράφεται αυτόματα, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να ζητήσει να τοποθετηθεί, να, να συμπεριληφθεί ένα θέμα ε, στη Μεσή Διάταξη και αποφασίζει ο πρόεδρος. Δηλαδή η διαφορά ποια είναι, ότι ενώ όλοι μπορούν να ζητήσουν, εδώ είναι σαφές ότι θα συμπεριλαμβάνεται ε, το θέμα αυτό στη Μεσή Διάταξη. Αν θέλουμε να αφαιρέσουμε αυτό το δικαίωμα, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός. Αν όμως αποφασίσουμε ότι ε, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες διευκρινήσεις, τότε πράγματι πρέπει να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε τον κανονισμό. Πάντως, η δική μου πρώτη αντίδραση είναι ότι πολύ δύσκολα μπορεί να υπάρχει μια ερμηνεία η οποία θα λέει διαφορετικά από αυτά που λέει ο κανονισμός. Αυτό υπάρχει σαν δικαίωμα των ε, βουλευτών, είτε αρέσει είτε όχι. Ε, δεν μπορούμε δηλαδή να δώσουμε μια αντιφατική ερμηνεία. Βεβαίως, ε, το θέμα αυτό δεν μπορεί να σημαίνει ότι το δικαίωμα αυτό υπερισχύει των άλλων δικαιωμάτων, δηλαδή αποτελεσματικότητα, ε, ο χρονισμός, το χρονικό σημείο. Ε, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προέχει, κατά την άποψή μου ακολουθεί. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, βρίσκεται στην ε, κρίση του καθενός, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δεν θέλουμε να διαγράψουμε, να αφαιρέσουμε αυτό το δικαίωμα, το οποίο έχουν σήμερα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Τρασκόφσκι. Συμφωνώ. για το 117. Αλλά αν αρχίσουμε συζήτηση επίσημη θα ανοίξουμε το κουτί μίας πανδόρης. Αυτό φοβάμαι, γιατί πολλά μέλη της ΑΦΕΤ θα το δεχτούν μεν, αλλά δεν θα διευκολύνει αυτό καθόλου τη δική μας δουλειά. Συνδέεται βέβαια και με άλλα θέματα, με τις γραπτές δηλώσεις, με συμφερόντων και άλλες πρωτοβουλίες που αφορούν τους βουλευτάς. Διότι νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν όλοι μαζί να το δούμε. Να μην συγκεντρώσουμε, να μην κεντρώσουμε την προσοχή μας μόνο σε αυτά τα δύο θέματα πέρα από την κανονική δουλειά του Κοινοβουλίου. Γιατί εδώ μιλάμε για πολλαπλά συμπτώματα της ίδιας ασθενείας. Πρέπει να τα δούμε κάποτε όλα μαζί και να μας απαντήσει η ΑΦΚΟ τι θέλει πράγματι. Γιατί όταν μιλάμε για τις γραπτές δηλώσεις και τις πρώτες αναγνώσεις έχουμε τέτοιες διχογνωμίες που δεν καταλήγουμε πουθενά. Πρέπει να επιμείνουμε στα θεσμικά, στις εκθέσεις ή προτάσεις ιδίας πρωτοβουλίας, στις δικαιοδοσίες μας ή σε θέματα που απλώς θα κάνουν μεγαλύτερη φασαρία. Είναι όλα αυτά συμπτώματα της ίδιας ασθενείας. Ο κύριος Ντάφ. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Το πρόβλημα τέθηκε για λόγο του φόρτου εργασίας της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, ε, Και ακόμη δεν ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει. Δεν έχει ακόμη οργανωθεί καταλήλως ώστε να μπορεί να απαντάει σε ερωτήσεις και μάλιστα εγκαίρως. Ελπίζουμε βέβαια αυτό να είναι προσωρινό το πρόβλημα και να μην διαιωνιστεί στις σχέσεις του Κοινοβουλίου με την υπηρεσία αυτή εξωτερικών διηράσεων. Δεν θα έπρεπε λοιπόν σε αυτήν τη φάση να θεσμοποιήσουμε τις διαφορές μας με την υπηρεσία αυτή αλλά να επιτρέψουμε στην υπηρεσία εξωτερικών δράσεων να τους δώσουμε λίγο χρόνο για να τα κανονίσει. Στην Επιτροπή Εξωτερικών υποθέτουν πάντοτε ότι τέτοια θέματα τελικά θα τεθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής. Δεν πρόκειται για καμία συνωμοσία του Προεδρείου. Ούτε προσπάθεια της ΕΠΕΚΣ να απαγώσει τα πράγματα. λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούμε προς το παρόν. Άρα σε αυτήν τη φάση θα ήθελα να επιδείξουμε μεγαλύτερο ρεαλισμό και να, αν όχι πραγματισμό καθαρά, και να πούμε ότι θα κάνουμε χρήση της κοινή λογικής και ότι αναγνωρίζουμε τη διακριτική ευχέρεια που πρέπει να έχει η υπηρεσία αυτή για να διακανονίσει τις εργασίες της. Αν τελικά αποδειχτώ υπερβολικά αισιόδοξο και σε κάνα δυο χρόνια συνεχίσει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τότε βεβαίως η ΑΦΚΟ θα έπρεπε να ξανασυζητήσει αυτό το θέμα και να ζητήσει μια πιο επίσημη αλλαγή στον κανονισμό. για να ζητήσει ας πούμε μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των βουλευτών ή μεγαλύτερη προστασία γενικότερα των βουλευτών. Αλλά επαναλαμβάνω δεν μου φαίνεται η καταλληλότερη χρονική στιγμή η τωρινή για να ζητήσουμε κάτι τέτοιο. Ας αφήσουμε μια περίοδο περισυλλογής και πραγματισμού. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να κάνω δύο διευκρινήσεις. Προηγουμένως, τελειώντας την παρέμβασή μου, είπα ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε ταχύτατα. Ε, ίσως όμως ε, καλύτερα να το αναβάλουμε για αύριο. Ε, δεν θα είμαι βέβαια εγώ παρόν, αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η πρώτη διευκρινήση. Η δεύτερη είναι η εξή. Στο κείμενο της ε, τροπολογίας που έχω καταθέσει, στην, ε, τροπολογία, στην γνωμοδότη στη δική μου, εκεί αναφέρεται ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει και ε, το δικαίωμα να ε, διαγράψει μια συγκεκριμένη, συγκεκριμένο θέμα από την ημερήσια διάταξη. Αλλά βέβαια πρέπει να συζητήσει με τον ε, άμεσα ενδιαφερόμενο. Το, η έννοια του άρθρου 117 νομίζω ότι είναι σαφής. Δεν λέει δηλαδή ότι στην πρώτη συνεδρίαση. Γιατί αν ας πούμε ε, η πρώτη συνεδρίαση είναι και την ημέρα που λύγει η προθεσμία, πώς θα γίνει αυτό. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως είναι σωστό. Αυτό που είναι το σωστό είναι να δώσουμε μία ρεαλιστική απάντηση, δηλαδή να αν δεν έχει δοθεί η απάντηση στον ερωτώντα, τότε μπορεί κανείς να μιλήσει στην Επιτροπή ε, για ε, το ποιο είναι το βέλτιστο και αυτό θα αποφασιστεί κοινού από τον εισηγητή και τον πρόεδρο. Και εγώ αυτό προτείνω και εσείς αύριο αν θέλετε υπερψηφίζετε ή καταψηφίζετε. Όπως σας είπα, αύριο δεν θα είμαι εδώ, γι' αυτό πρέπει να τα πω όλα σήμερα υπάρχει βέβαια και η έκθεση Ταρκόφσκη, ας ελπίσουμε να τη συζητήσουμε και αυτό. Τώρα, η επόμενη δική μου έκθεση αφορά τον, ε, την τροποποίηση των άρθρων που αφορούν την τροποποίηση των άρθρων 87α 88 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα παλιά 290 και 291 σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ε, ξέρετε πολύ καλά, έχει ε, επικαιροποιηθεί ε, το η διαδικασία της επιτροπολογίας. Νομίζω όμως ότι τα έχουμε πει όλα αυτά ε, και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Εγώ απλά πρέπει να ε, τοποθετηθώ σε αυτά τα δύο θέματα και εσείς ε, να στηρίξετε τις δικές σας τις τροπολογίες γιατί κατατέθηκαν αρκετές τροπολογίες. Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι νομοθετικές διατάξεις που αναθέτουν στην Επιτροπή να εξετάσει θέματα μέσα σε ορισμένα χρονικά πλαίσια, εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, να ζητήσει τροποποιήσεις ή να εγκρίνει. Εν πάση αυτά βρίσκονται υπό τον ε, έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το Κοινοβούλιο μπορεί και να ανακαλέσει την εντολή που έχει δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ το παλιό άρθρο αναφέρεται σε εκτελεστικές πράξεις ε, και στην περίπτωση αυτή πράγματι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση του ελέγχου. Το σχέδιο της έκθεσης ε, το οποίο προτείνω εγώ θέλει να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες κυρίως για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και γίνεται ιδιαίτερος, ιδιαίτερη μνήα για την ε, ε, δυνατότητα ε, γίνεται ιδιαίτερη μνημεία στις εκτελεστικές πράξεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται, όπως σας είπα, εξέταση εκτελεστικών στην περίπτωση αυτή μπορεί κανείς να ζητήσει την ανάκληση των προτάσεων της Επιτροπής με βάση την Γενική Αρχή ότι ακόμα και αν υπάρχει ειδική αρμοδιότητα της ε, Επιτροπής ε, της Αρμόδιας επιτσουσίας δεν μπορεί κανείς ε, να αφαιρέσει από το Κοινοβούλιο την δυνατότητα να παρεμβαίνει <laughs> βεβαίως μετά από αίτημα που θα υποβληθεί ε, από 40 βουλευτές ή και από περισσότερους. Ε, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να επιταχύνεται η όλη διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα ε, να τεθούν ταχύτατα σε ισχύ τα, οι εκτελεστικές πράξεις. Εγώ σε γενικές γραμμές ε, συμφωνώ βέβαια ε, με εκείνους ε, που επιθυμούν τον συμβιβασμό. Μπορούμε παραδείγματο χάρη να πούμε ότι οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από μπορούν πράγματι να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο ενός συμβασμού. Η τροπο τροπολογία υπαριθμών 5. Εκεί αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αναφέρεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ε, σε όλα τα θέματα ή ε, όταν υπάρχει το θέμα του συμβασμού, το πρόβλημα που τίθεται είναι ε, κατά πόσο είναι αρμόδια για τις ε, κατεξοδότηση πράξη μια συγκεκριμένη επιτροπή. Όσον αφορά τις ε, άλλες τροπολογίες, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, μεγάλες ε, διαφορές σε σχέση με αυτά που πρότεινα. Παραδείγματο χάρη, η ιδέα, αυτά που είπε ο συνάδελφος Νταφ, δηλαδή της κατεξουδότηση πράξης να τις παραπέμψουμε σε μια συγκεκριμένη επιτροπή, αυτό κατά την άποψή μου είναι μια γραφειοκρατική παράταση. Ε, αναφέρεται ότι οι αρμόδιες επιτροπές θα πρέπει να λαμβάνουν τις κατεξοδότηση πράξεις. Πρόκειται για την τροπολογία υπαριθμών 21 του κυρίου Νταφ άλλοι αναφέρονται στην διάσκεψη των Προέδρων. Νομίζω ότι επ' αυτό έχω ήδη τοποθετηθεί. Η τροπολογία Μερέιρα, αν κατάλαβα καλά, εκεί προτείνεται ε, να ε, περιμένει κανείς ε, να εκπνεύσει το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για τις παρεμβάσεις της Επιτροπής. Και εγώ νομίζω όμως ότι το χρονικό διάστημα ξεκινάει από τη στιγμή που έχουν διανεμηθεί οι μεταφράσεις των γραπτών κειμένων. Αυτό μπορεί να είναι λεπτομέρεια, αλλά νομίζω ότι μπορεί κανείς να το αναφέρει. Σε άλλες πάλι τροπολογίες ε, γίνεται λόγος ε, για, τους, ε, για τα αίτια των αντιρρήσεων. Πάντως θεωρώ ότι δεν πρέπει κανείς να περιορίζει την συνθήκη της Λισαβόνας, να περιορίζει αυτά τα οποία αναφέρει η συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Και ε, υπάρχουν και άλλες ε, τροπολογίες που μπορούν να συζητηθούν, που έχουν ως στόχο γενικότερες ε, απόψεις και όχι ιδιαίτερες ε, λεπτομέρειες. Οι τροπολογίες 35 και 37, οι τροπολογίες αυτές ε, μοιάζουν, αλλά παραδείγματο χάρη η τροπολογία υπαριθμών 35 διευκρινίζει... Μισό λεπτό. Νομίζω ότι είναι η τροπολογία του κυρίου Μορέιρα. Με αυτή την τροπολογία αποκλείονται από την κατάσταση τροπολογιών οι μη γεγραμμένοι. Η, η τροπολογία Βέμπερ, η 37, ε, Άλλες τροπολογίες, ε, η 47 του Ντάφ, η 48 του Μορέδα, η 38 του Μορέδα, η 39 του Μορέδα, αυτές μπορώ να τις συμπεριλάβω. Νομίζω τώρα βέβαια δεν πρέπει να εξετάσουμε κάθε μία τροπολογία μεμονωμένα. Εγώ νομίζω ότι εκείνο που είναι σημαντικό είναι να μην επιβαρύνουμε, να μην ε, καταστήσουμε ακόμα πιο δυσκίνητη μία διαδικασία όπου προβλέπεται ότι πέρα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκεί το κοινοβούλιο και που είναι απαραίτητο, θα πρέπει ε, να υπάρχει και μία, ε, ένας συγκεκριμένος αριθμός, μία ταχύτητα στην εξέταση των διαδικασιών. Ε, βεβαίως, ε, ε, οι συνάδελφοι μπορούν να πούν την άποψή τους και η ψηφορία θα γίνει σε άλλη περίπτωση. Ο κύριος Νταφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αλλά και σημαντικό το θέμα αυτό. Και θα πρέπει το Κοινοβούλιο αποτελεσματικά να προσαρμοστεί στο νέο καθεστώς με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μέχρι στιγμής υποπτεύομαι ότι ήταν λίγο ασαφής η κατάσταση σε κάποιες επιτροπές ως προς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν σε ό,τι αφορά τις ε, κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικέ πράξει. Πολύ σωστά είπατε ότι εξέτασα λίγο αυτό το ενδεχόμενο επιτροπή κάποιων ειδικών εμπειρογνωμόνων υπαλλήλων οι οποίοι θα αποπτεύονταν από τους βουλευτές και θα έκανε ουσιαστικά το πρώτο που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, να δίνουν ε, τις πράξεις στην αρμόδια, κάστοτε αρμόδια επιτροπή. Αλλά σε αυτή την ε, παράδοση θα έπρεπε να αναφέρουν και το βαθμό της σοβαρότητας και του κατεπήγοντος και να δίνουν προτεραιότητα σε κάποια σημεία προς την ε, Επιτροπή, την αρμόδια, τα σημεία εκείνα τα οποία έχουν πολιτική σημασία, δηλαδή θα έπρεπε να τα προβάλλουν. Η πρόταση ως έχει αυτή λέει ότι η Προεδρία διαδίδει απλά με ουδέτερο τρόπο, χωρίς σχόλια δηλαδή, τις πράξεις της εκάστοτε αρμόδιες επιτροπές και εγώ θα έλεγα ότι καλό θα ήταν μια πιο εξειδικευμένη επιτροπή να είναι αυτή η οποία θα μπορούσε έτσι να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια. Αν όμως εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι γραφειοκρατικό και χρονοβόρο, τότε θα αποσύρω αυτή την ιδέα. Να πω και κάτι άλλο. Έχω καταθέσει την τροπολογία υπερθμών 29, στην οποία λέω ότι ευκταίο θα ήταν στην Ολομέλεια ο Πρόεδρος να θεσπίζει μία περίοδο που θα αφήνει πλέον εκτός οποιαδήποτε περιθώρια αμφιβολίας. Αν δηλαδή ανακοινώνεται ένα χρονοδιάγραμμα, μπορεί αυτό να βοηθήσει το έργο των επιτροπών. Σε ό,τι αφορά τώρα την τροπολογία 35. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω το ζήτημα των ε, συνόδων της ε, Ολομέλειας στις Βρυξέλλες. Που αρχικά δεν συμπεριλαμβάνονται στην τροπολογία 4, στην αρχική διατύπωση. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε αυτό το πρόγραμμα, το προπαρασκευαστικό των ε, Ολομελιών των Βρυξελών, που είναι πιο σφιχτό διάγραμμα και να έχουμε μια σαφή αναφορά σε ό,τι αφορά τις και κατεξουσιοδότηση πράξη. Πέραν αυτού όμως, φαντάζομαι ότι όλοι συμμεριζόμαστε το πνεύμα των προτάσεών σας και είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να καταλήξουμε τελικά σε μια καλή συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όλες οι προτάσεις τροπολογιών στόχο έχουν τη διευκόλυνση και την ταχύτερη δεκπεραίωση της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου για τις κατεξουσιοδότης συμπράξεις και για τις εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ νομίζω ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να το αναλάβει αποκλειστικά η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Στην εκάστοτε περίπτωση και όταν είναι πάνω από μία, αυτές. Και μόνο στην τελική απόφαση θα πρέπει να παρεμβαίνει η Ολομέλεια. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να παρεμβαίνουν οι πρόεδροι των επιτροπών, μόνο αν υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ δύο περισσότερων επιτροπών. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε κάτι που δεν έχουμε πετύχει πάντοτε. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την, τον πολλαπλασιασμό των ειδικών διαδικασιών που είναι πολύπλοκες, μακροσκελείς, χρονοβόρες διαδικασίες. Διότι ποιος είναι ο κίνδυνος. να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο και προσπάθεια και οι βουλευτές των Επιτροπών και οι πρόεδροι των Επιτροπών και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Και ο πρόεδρος της διάσκεψης των πρόεδρων των Επιτροπών. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και γι' αυτό θεωρώ ότι θα έπρεπε να ασχοληθούμε πολύ σοβαρότερα και περισσότεροι να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Είμαστε νομοθετικό σώμα, άρα εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε τις εργασίες μας. Με ανησυχεί αυτή η πρόταση για τη δημιουργία ενός συνόλου μηχανισμών που απαιτούν τόσο χρόνο, τόσο μεγάλες προσπάθειες που τελικά θέτει σε κίνδυνο την άσκηση του βασικού μας καθήκοντος, του νομοθετικού καθήκοντος. δεν έχουμε μόνο το θέμα τη ε, δημοκρατική νομιμότητα και νομιμοποίηση που πρέπει να μας απασχολεί, αλλά θα πρέπει να δούμε και αν μπορούμε, να είμαστε σε θέση να εφαρμόζουμε με επαρκή τρόπο να εκτελούμε τις αρμοδιότητές μα. το deliver, δηλαδή να παραδίδουμε αποτελέσματα. Πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και αποδοτικοί. Να πούμε στους συμπολίτε μας ότι ακούστε τον χρόνο σας και τους πόρους τους αξιοποιούμε, τους χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είμαστε ικανοί να φέρουμε σε πέρα το λειτουργήμά μας, ε, ε, πέρα στο λειτουργήμά μας, να ασχίσουμε τις ε, αρμοδιότητές μας. Και σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχουν καθυστερήσει για μήνε ό,τι αφορά τι εκτελεστικέ πράξει ή τι κατεξουσιοδότηση πράξη. Γιατί μια τέτοια καθυστέρηση θα μπορούσε να συνεπάγεται και προβλήματα για την Ένωση γενικά. Δηλαδή λέμε στην Κομισιό να <clears throat> προτείνει, να εφαρμόσει κάποιες προτάσεις και μετά ξαναρχίζουμε να εξετάζουμε τα πάντα και καθυστερούμε ολόκληρους μήνες. πρέπει να είμαστε κάπως ε, συνεπείς. Τι θέλουμε τελικά. Θέλουμε η Κομισιόν να είναι αυτή η οποία μέσω των κατεξουσιοδότηση πράξεων να κάνει αυτά το οποία εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε υπό καλύτερες συνθήκες. Και αν ναι, τότε γιατί στη φάση του ελέγχου κατόπιν. Ενεργούμε ως ε, εκτελεστικό σώμα. Πρέπει ε, να είμαστε πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί, επαναλαμβάνω, στις εργασίες μας. Κύριε Σάγνιο, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Τι να σας πω, δεν θα ήταν καλύτερο την πηγή αυτού του προβλήματος να την αντιμετωπίσουμε δηλαδή. Να καλέσουμε την ε, Βαρόνη Άστον. Αυτό κάνουν τα πραγματικά κοινοβούλια. Έχει ένα τεράστιο μισθό. Πάρα πολλά χρήματα δαπανά το τμήμα τη, η υπηρεσία τη, έχει πάρα πολύ προσωπικό και παρόλα αυτά αδυνατή εγκαίρω να απαντήσει όλα αυτά τα ερωτήματα. Αυτό πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε και όχι πώ θα συγκαλύπτουμε κάποια γεγονότα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Ε, δεν βλέπω να έχει στήσει κανείς άλλο το λόγο. Κατόπιν τούτου, ε, νομίζω ότι υπάρχει ε, συνένεση, αν θέλετε, όσον αφορά το σχέδιο της έκθεσης το οποίο σας παρουσίασα. Ο συνάδελφος κύριος Νταφ επέμεινε σε ορισμένα θέματα, αλλά είπε επίση ότι είναι και πρόθυμος ε, να συζητήσει και να ζητήσει τον συμβασμό. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Μορέιρα, ε, θέλω να πω το ότι εδώ υπάρχει αυτή όλη η ιδέα του να προκύψει επιτάχυνση. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να οριστεί η μερομηνία των ψηφοφοριών το Μάρτιο κάποια στιγμή. Και στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα θα δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρξουν και κάποιοι, να κάποιο συμβασμό. Δεν βλέπω να είμαστε πολύ μακριά ε, στις απόψεις μας, αλλά αν υπάρχει κάποια δυνατότητα συμβασμού, γιατί όχι. Ας ε, καταλήξουμε λοιπόν ε, σε αυτό, να ψηφίσουμε το Μάρτιο. λοιπόν, εγώ τις δικέ μου τις εκθέσεις τις είπα όλες, τα εξάντλησα και τώρα θα ήθελα μισό λεπτό διακόπτη πρόεδρος. Sì, sì, sì, certo, abbiamo ancora tempo e anzi siamo in anticipo io ho chiesto Έχουμε κερδίσει χρόνο εγώ είπα να ξεκινήσει συνεδρίες των συντονιστών στις 5 και τώρα είναι 4 και 5 έχουμε όσο χρόνο θέλετε για να ασχοληθούμε με την έκθεση Ταρκόφσκι με την 7 λοιπόν που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 123 του κανονισμού ε, που αφορά στις γραπτές δηλώσεις. Ο κύριος Τσαρκόφσκι είναι ο εισηγητής, τον ορίσαμε πέρυσι το Φεβρουάριο και τον παρακαλέσαμε να μελετήσει ε, το θέμα αυτό το έκανε και σας ε, με τις απόψεις του. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ταρκόφσκι ε, να ε, μας ε, πει τις δικές του τις απόψεις σχετικά με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Για τις γραπτές δηλώσεις. Σε μια προηγούμενη ζωή ήμουν καθηγητής και γι' αυτό Ζήτησα να γίνει μελέτη για αυτές τις δηλώσεις συμφερόντων για να δω αν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Αν δηλαδή βελτιώνεται η νομοθετική διαδικασία με αυτές ή αν μήπως είναι απλώς μια περίπτωση δημοσίων σχέσεων. Δυστυχώς είχα δίκιο τελικά σε αυτά που υποπτευόμουν. Οι γραπτές δηλώσεις δεν επηρεάζουν, δεν βελτιώνουν την νομοθετική διαδικασία. Απευθύνονται στην Κομισιόν, η οποία μετά μας πληροφορεί απλώς ότι κάτι έκανε ως αντίδραση. Το αποτέλεσμα είναι πολύ περιορισμένο. Οι συντάκτες της έκθεσης δεν κατάφεραν να ονοματίσουν κανένα παράδειγμα βελτίωσης της νομοθετικής διαδικασίας με τις γραπτές δηλώσεις. Με βάση εκατοντάδες από αυτές. Και τώρα θα αναφέρω ορισμένους κανόνες που πρέπει να θεσπίσουμε, μα ζητούν να θεσπίσουμε. Αλλά πρώτα να δούμε πώς έχει η κατάσταση με τις γραπτές δηλώσεις και αν τις χρειαζόμαστε. Από τη μία λοιπόν έχουμε τώρα τις δικαιοδοσίες που έχουμε και δεν έχουν πια πολύ νόημα οι γραπτές διαδικασίες αυτές οι δηλώσεις. Είχε, ήταν της εποχής όπου το κοινοβούλιο δεν είχε τόσες δικαιοδοσίες και τώρα έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από την Κομισιόν να αναλάβει πρωτοβουλία. Άρα οι γραπτές αυτές δηλώσεις δεν είναι πολύ αποτελεσματικές. Απ' την άλλη όμως καμιά φορά μας λένε οι συνάδελφοι ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να τεθεί κάποιο θέμα που είναι σημαντικό για τους εκλογείς των Άλλοι λένε ότι για μερικούς βουλευτές δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ξεκινήσει μια νομοθετική διαδικασία και να προσεχτεί έτσι κάποιο πρόβλημα που τους ενδιαφέρει. Έχετε όμως δει πόσες υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις και οι περισσότερες δεν έχουν νόημα. Αυτή ήταν η εισαγωγή. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαρχαιωμένο εργαλείο δεν έχει καν χρησιμοποιηθεί πολύ και δεν είναι σωστό να λέμε ότι είναι σημαντικό, αν και για μερικούς βουλευτές μπορεί να έχει περισσότερη σημασία. Τι προτείνω λοιπόν. Θα δούμε πρώτα ποια είναι τα συμπεράσματα της μελέτης. Δεν είναι, λέω, εργαλείο πολύ αποτελεσματικό και έχει απαρχαιωθεί μετά από τις διαδικασίες που έχουμε τις καινούργιες τώρα. Τέλος λέω ότι στην επόμενη θητεία πρέπει να σκεφτούμε και το μέλλον τους αυτών των δηλώσεων. Δεν προτείνω μεν καμία συγκεκριμένη λύση, αλλά, αλλά να. Θα δείτε στο κείμενό μου ότι έχω κάποια άποψη. Βασικά λοιπόν δεν προτείνω καμία δραστική αντίδραση, αλλά στο μέλλον να το δούμε. Τώρα για τις λεπτομέρειες. θα ήθελα οι κανόνες για αυτές τις γραπτές δηλώσεις να είναι πιο συγκεκριμένοι τον αριθμό των υπογραφών, πότε μπορούν να αποσυρθούν κλπ. Βάζω λοιπόν μια διαφορετική διατύπωση και λέω ότι οι γραπτές δηλώσεις πρέπει να θίγουν θέματα για τα οποία έχει δικαιοδοσία η Ένωση. Και το λέμε αυτό πιο έντονα. Επίσης θέτω το σημαντικό θέμα να μην επικαλύπτονται με την υπόλοιπη νομοθετική διαδικασία, αυτό το λέει ήδη. Αλλά προσδιορίζω ότι πρέπει να έχουν σχέση με την κοινοβουλευτική δουλειά και να μην υπάρχει επικάλυψη με τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας ας πούμε. Ύστερα με κάποιον περισσότερο εξυγχρονισμό να δημοσιεύονται στο ίντερνετ, στο εσωτερικό του κοινοβουλίου και να διαδίδονται και με άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους. Να μπορεί κανείς δηλαδή να δει τον κατάλογο τους στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για τις υπογραφές. Οι υπογραφές πρέπει να μπορούν να αποσύρονται μέσα σε τρεις μήνες από την ε, συλλογή τους και εδώ το σημαντικό είναι μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες, αυτοί οι τρεις μήνες να είναι η διορία και όχι παραπάνω. Γιατί αλλιώς θα υπάρχουν δύο προβλήματα. Ένα, ότι οι συνάδελφοι απέσυραν τις υπογραφές τους όπως ήθελαν και όποτε ήθελαν, αφού είχε κατατεθεί μία και συμφωνηθεί μία δήλωση. Και έτσι αυξανόταν η σύγχυση αν θέλει λοιπόν κανείς να αποσύρει την υπογραφή του, να σέβεται την τρίμηνη διορία. Έπειτα μερικές φορές υπήρχε παράταση για την συλλογή ήδη των υπογραφών και αυτό νομίζω πρέπει να καταργηθεί. Για να συνοψίσω λοιπόν. Το θέμα των γραπτών δηλώσεων το αφήνω ανοιχτό γιατί είναι πολύ αμφιλεγόμενο. Θα ήθελα να επιδείξουμε κάποια μεγαλύτερη φιλοδοξία όμως και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τις καταργήσουμε. Το αφήνω πάντως ανοιχτό. Υπάρχουν και θέματα που αφορούν το πώς θα συλλέγονται οι υπογραφές και η κυρία Λούλινγκ το επεξεργάζεται αυτό Νομίζω ότι το ίντερνετ θα μας βοηθήσει πολύ και θα κάνει τη διαδικασία πιο διαφανή. Όσο δε για τους κανόνες εφαρμογής αυτού του εργαλείου να είναι σαφέστεροι, πιο συνεπείς και να καταφέρουμε μόνο οι γραπτές δηλώσεις που τις υποστηρίζουν πράγματι οι συνάδελφοι να γίνονται δεκτές. Γι' αυτό έβαλα αυτή τη τρίμηνη διορία για τις αποσύρσεις για να είμαστε λίγο αυστηρότεροι ως προς το χρόνο που διαθέτουμε για τις αποσύρσεις. Ευχαριστώ. Γκουρμάι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά πάντοτε συνεργάζομαι με τον Ραφαέλ και θα ήθελα να μιλήσω και για αυτή τη μελέτη του τμήματος ε, πολιτικής που να μας δώσει μια πολύ καλή επισκόπηση. Δεν είμαι κατά επί της αρχής των γραπτών δηλώσεων, αλλά είναι καλό για να εκφράζουν τις, ειδικές, τις ιδιαίτερες ανησυχίες τους οι βουλευτές. Σίγουρα έχουν και άλλα βέβαια μέσα ε, στη διάθεση για να το πράξουν αυτό. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των γραπτών δηλώσεων, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί σημαντικά. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι τα μέλη, οι βουλευτέ γνωρίζουν πια το εργαλείο αυτό και έχουν κάποιες ιδέες για το πώς μπορούν να εξοπλίσουν ακόμη περισσότερο ε, και με πιο σοφό, θα έλεγα, τρόπο αυτό το θέμα, επειδή ε, το θέμα μπορεί να τους ενδιαφέρει αντικατοπτρίζουν και απόψει των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό δεν είμαι υπέρ τη κατάργηση των γραπτών δηλώσεων, αλλά υπέρ τη μεταρρύθμιση αυτής της διαδικασίας. Είμαι υπέρ του να υπάρχει μια αποκλειστική online πλατφόρμα για γραπτές δηλώσεις, ε, γιατί πλέον έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και η τεχνολογία. Επίσης δεν χρειάζεται να δαπανούμε τόσους πόρους σε χαρτί. Να μην παρατείνουμε την ε, τριμήνη περίοδο επίσης, πιστεύω. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η δημοσιότητα, η δημοσιοποίηση αυτών των γραπτών πρέπει να είναι περιορισμένη. γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχει ε, άσκηση πίεσης μπροστά από το ημικύκλιο, με πόστρηση οτιδήποτε άλλο αλλά σε, ε, μεταξύ των θεμάτων των γραπτών δηλώσεων θα μπορούσε να περιλαμβάνονται οι τρέχουσες νομοθετικές διαδικασίες. Έχουμε δει να μην συγκεντρώνονται υπογραφέ αρκετέ για κάποια θέματα. Αλλά έχουμε δει και επιτυχημένε γραπτέ δηλώσει. Αν υπάρχουν κάποια κριτήρια, ίσως ε, ο παραλήπτης θα μπορούσε να απαντά αν υπάρχουν δηλαδή σε αυτή τη δήλωση κάποιες ομάδες που προσωπούνται, ως ιδέα το αναφέρω. Δεν είμαι απόλυτα βέβαια για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. Πάντως θα συνεργαστούμε, πιστεύω πολύ καλά και θα έχουμε κάτι καλό. Σίγουρα καλό είναι να μην στερηθούμε αυτό το εργαλείο, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ένα είδο πρωτοβουλία των πολιτών, αλλά πρωτοβουλία θα έλεγα των Ευρωβουλευτών. Κρίνει ο συγκεκριτή ε, τη γραπτής λύση με βάση δύο κριτήρια. Το αν καθορίζουν την ατζέντα των θεσμικών οργάνων και το αν επηρεάζουν τελικά τι ε, αποφάσει που λαμβάνονται. Και στι δύο ερωτήσει, νομίζω ότι σαφής είναι απάντηση. Είναι όχι. Άρα αυτά τα δύο κριτήρια πρέπει να τα ε, καταρρύψουμε. Δεν τα δέχομαι. Η πολιτική τάξη του Κοινοβουλίου είναι αυτή η οποία ορίζει την ημερήσια διάταξη και εδώ και αντίστοιχα και στα άλλα θεσμικά όργανα. Και αυτή η πολιτική τάξη λαμβάνει και τις αποφάσεις. Τώρα, για θέματα που δεν πρόκειται να μπουν ε, στη ημερήσια διάταξη, αν έχουμε κάποιες ε, ε, απόψεις μειοψηφίας ε, κάποιων βουλευτών, δεν ξέρω. Ίσως χάνουμε το χρόνο μας κάποιοι από εμάς, αλλά Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ε, χάσιμο χρόνο το να εκφράζει κανείς ε, την άποψή του, ακόμη και αν είναι στην μειοψηφία, μάλλον ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και μάλιστα βλέπουμε ότι κάποιες αποφάσεις ε, πολύ σημαντικές, όπως κατάρρηση της δουλείας, η ε, μεταρρύθμιση των ε, εργασιακών συνθήκων ε, μπορεί να διαβάσει την ιστορία και να δει πώς εξελίχθηκαν. Ίσως ξεκίνησαν από κάποια μειοψηφία. Υπάρχουν κάποιες απόψεις που μπορεί να εκπροσωπούνται από μια μειοψηφία, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δημοσιοποιηθούν παρόλα αυτά. Έχουμε διάφορα θέματα κάποιους Βρετανούς κτηνοτρόφους, Ισπανούς ε, που διαμαρτύρονται για την αναρχιδόμηση ακτές και ούτω καθεξής, ή κάποια σκυλιά μπορεί να κανένα. Μπορεί κάποιος να θεωρούν αυτά τετριμένα θέματα, αλλά είναι σημαντικό να αναφέρονται. Well, I, um, Δεν το έχω ακόμη συζητήσει με την ομάδα μου το θέμα αυτό για να δούμε τι άποψη επικρατεί. Είναι πάντως πάρα πολύ δημοφιλής, περιέργως θα έλεγα, οι γραπτές δηλώσεις και αν η Επιτροπή αποφασίσει την κατάργησή τους, ίσως γίνουμε στόχος μεγάλης κριτικής. Γενικώ στο σώμα. αλλά φαντάζομαι ότι και η δημόσια κοινή γνώμη θα μας κρίνει. Η οργανωμένη κοινότητα των πολιτών, κυβερνητικέ οργανώσεις. Συχνά προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτές τις γραπτές δηλώσεις. Και είναι κάτι που τους αρέσει. Κάποιε φορέ προτιμούν να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίε εσωτερικά μέσα στο Κοινοβούλιο, μέσα από αυτή τη διαδικασία των γραπτών δηλώσεων και όχι να ξεκινήσει με κάποια εξωτερική πίεση. Κάποιοι βουλευτέ μπορούν επίσης να εκφράσουν την ανεξαρτησία του από την υπόλοιπη ομάδα τους. να συμπήξουν συμμαχίες μέτωπα ανεξαρτήτως πολιτικής ε, κομματικής πειθαρχία, ε, άτομα τα οποία ε, έχουν την ίδια άποψη για κάποιο θέμα. Και αυτό το δικαίωμα το δίνει, αυτή τη δυνατότητα τη δίνει αυτή τη δικασία των δηλώσεων στους βουλευτές. Και μου αρέσει αυτή η προσέγγιση η διακομματική, υπερκομματική, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι. <laughs> Πάντως θεωρώ ότι όταν ο πρόεδρος ασκεί τη δεκτική του ευχέρεια, κατά περίπτωση, βάσει τον ισχύοντα κανόνα, θα μπορούσε να ασκεί μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια με ένα ποιοτικό έλεγχο. Και πιστεύω ότι κάποιες από τις πρόσφατες γραπτές δηλώσεις δεν ε, είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάπως τα υπερβαίνουν και θα πρέπει να μπαίνουν κάποια κριτήρια να δούμε και ποια είναι η δυνατότητα που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι πρωτοβουλίε μπορεί να αναλάβει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε να επιδείξουμε κάποια αυτοσυγκράτηση στι ε, γραπτέ ε, δηλώσει, αλλά θα μπορούσαμε να στείλουμε σε εξωτερικού ε, το λάθο μήνυμα, αν δεν την επιδείξουμε την αυτοσυγκράτηση, <clears throat> ότι έχουμε μεγαλύτερε εξουσίε από αυτέ που πραγματικά έχουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, Εγώ νομίζω ότι μπορούμε και είναι ε, σκόπιμο να μπορούμε να εκφράζουμε την άποψή μας για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος. Όπως ε, Συμβούλιο της Ευρώπης, για παράδειγμα. Πρόσφατα υποστήριξα μία προσπάθεια επέκτασης του franchise σε άτομα με αναπηρία. Δεν είναι ακριβώς αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι ένα θέμα που σίγουρα ξεκάθαρα ενδιαφέρει τη δημόσια κοινωνία. Και νομίζω ότι είναι ένα τομέα που περιμένει από εμά να αναλάβουμε δράση, Είναι κοινή γνώμη. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια δύσκολη ισορροπία, δεν είναι εύκολο. Δεν είμαι σίγουρη ότι επιτυγχάνεται αυτή η ισορροπία με τον κανόνα όπω ισχύει αυτή τη στιγμή. Τόσο διαφορά τις μη νομοθετικές διαδικασίες και την τροπολογία σας, δεν ξέρω. Τι εννοείται ακριβώ. Εκθέσει ειδήσει πρωτοβουλία τη Επιτροπή Εξωτερικών περιλαμβάνονται. για κάποια, παραδείγματο χάρη, υπόθεση διεθνή όπω είναι το Παλαιστινιακό ή η πυρηνική ανάπτυξη πυρηνικών ε, στο Ιράν. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα θα είναι να σταθμίσω θα υπέρ και τα κατά να διαβουλευτώ και με την ομάδα μου που κάποιες φορές ε, βοηθά, με βοηθά και εμένα να μορφώσω άποψη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εξετάστε το ενδεχόμενο να περιορίσετε τον αριθμό των γραπτών δηλώσεων. Για μια συγκεκριμένη μιλάμε χρονική στιγμή. Γιατί αν υπάρχει πολλαπλασιασμός σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή αυτών των δηλώσεων ε, υποβαθμίζει την πολιτική σημασία μιας συγκεκριμένης ε, δήλωσης. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή όχι μόνο το σκέλος της ποιότητας αλλά και της ποσότητας. An MEP with a good idea could um, put a bid in. Και ίσως θα πρέπει να ορίσουμε κάποιες ποσοστώσεις, ενδεχομένω. Ετησίως. Να υπάρχουν δηλαδή κάποια νότατα όρια. που θα εντάξουμε σε αυτό το μηχανισμό των γραπτών δηλώσεων. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Πριν λοιπόν δώσω τον ε, λόγο ε, σε άλλου, ε, θα μου να δώσω λόγο στον κύριο Χέφνερ. Κοιτάξτε μου, μία σύντομη ερώτηση. Καταρχήν, δεν θέλω να περτώ σε κάτι το οποίο προς το τέλος είπε ο κύριος Άντριου Νταφ, δηλαδή και εγώ επιθυμώ το όλο θέμα αυτό να το εξετάσω με την ησυχία μου και να το συζητήσω στην πολιτική μου ομάδα. Γιατί ε, το πρόβλημα με τις ε, γραπτές δηλώσεις ε, είναι ο πληθωρισμός που συνεπάγεται. Τόσο όσον αφορά την σημασία του, όσο και την ποιότητα. Κατόπιν τούτου, αυτό που, έχει, που νομίζω είναι σημαντικό είναι να βρεθούν εργαλεία τα οποία θα προκαλούν καλύτερη ποιότητα χωρίς ε, να προκύπτει αποδυνάμωση. Επιτρέψτε μου όμως τώρα πολύ σύντομα να αναφερθώ ε, στο θέμα αυτό το οποίο συζητάμε ε, σήμερα. Και θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω κατά πόσον ενδεχομένως με την εφαρμογή του άρθρου 177 του καταστατικού μας ε, κατά πόσον υπάρχει το δικαίωμα ανα πάσα ώρα και στιγμή ένα μέλος της Επιτροπής να ζητήσει την αναβολή εξέτασης του θέματος ή να αφαιρεθεί το θέμα από την ημερήσια διάταξη. Με βάση λοιπόν ε, τον ε, κανονισμό 114 7 παράγραφος 3 ένα θέμα πράγματι εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη, αλλά αν ε, κρίνεται ότι δεν ενδείκνεται το θέμα αυτό να συζητηθεί τη συγκεκριμένη μέρα, τότε νομίζω ότι η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει για μετάθεση εγγραφής του θέματος στην ημερήσια διάταξη. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ταρκόφσκι, ε, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ε, θέλω να πω ότι όταν πάμε στην Ολομέλεια, δεν το κρύβω αυτό, ε, μας περιβάλλουν οι ομάδες πίεσης και αυτό κατά την άποψή μου δίνει μια κάπως φεδρή εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Το δεύτερο που πρέπει να εξετάσει κανείς είναι το εξής. Πολύ συχνά οι συνάδελφοι υπογράφουν ε, χωρίς καν να διαβάσουν τη δήλωση. Τους παρασύρουν, τους λένε υπόγραψε και υπογράφουν αυτοί. Αυτό όμως δεν είναι σοβαρό, γιατί ε, πρέπει κανείς να προσέχει τι ακριβώς υπογράφει. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι οι γραπτές δηλώσεις, τουλάχιστον στην ε, ψυχολογία του ε, Ευρωπαϊκού του Ευρωβουλευτού, αντικαθιστούν λιγάκι αυτή την ε, γνωμοδότηση που υπάρχει. Αν ένας βουλευτής επιθυμεί να γίνει γνωστός, προετοιμάζει ένα νομοσχέδιο. Δυστυχώς όμως εμείς δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα ανάλυση πρωτοβουλίας. Και αυτό αντικαθίσταται από μία δήλωση. Βεβαίως, για να μπορεί κανείς να καταθέσει ε, μία γνωμοδότηση, ε, θα έπρεπε να έχει συγκεκριμένα δικαιώματα, θα έπρεπε να αλλάξει λιγάκι ο κανονισμός του Κοινοβουλίου. Εγώ πάντως θεωρώ ότι πρέπει να απαλλαγούμε από όλο αυτό το folklore, ε, το οποίο αφαιρεί από τη σοβαρότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Ταρκόφσκι, ο κύριος Κουαλτιέρη θέλει να πει κάτι. Θέλω μόνο να ε, τοποθετηθώ σε αυτά που μόλις τώρα είπατε και που τα κρίνω πολύ σωστά. Κοιτάξτε, όπως ε, ήδη ανέφερε η συνάδελφος ε, κυρία Γκουρμάη και συμφωνώ λιγάκι και με αυτά που είπε ο κύριος Ταρκόφσκι, Νομίζω ότι πράγματι θα πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι το πώς μπορούμε να οδηγήσουμε τους βουλευτές να έρχονται περισσότερο σε επαφή μεταξύ τους, κυρίως όσον αφορά το άρθρο 127. Είναι ένα άρθρο της συνθήκης, το οποίο κατά κάποιον τρόπο ε, προσχεδιάζει το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επειδή λοιπόν αυτό το Κοινοβούλιο γίνεται όλο και περισσότερο νομοθετικό ε, και σε θέματα προϋπολογισμού και σε θέματα πολιτικά. Πιστεύω λοιπόν ότι οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να εξελίσσονται με βάση αυτά, αυτούς τους στόχους που σας ανέφερα. Το θέμα δεν είναι να περιορίσουμε το δικαίωμα των ευρωβουλευτών να έχουν τη δική τους την άποψη, αλλά σιγά σιγά να μεταβιβαστεί ε, αυτό το θέμα των γραπτών δηλώσεων σε άλλο επίπεδο, Το που έχει σημασία είναι να μπορεί κανείς να ορίσει την ημερήσια διάταξη. Κυρίως όσον αφορά ε, εκθέσεις πρωτοβουλίας, εκθέσεις οι οποίες ε, καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απλά έτσι σκέφτηκα δυνατά για το πώς μπορούμε να δώσουμε μια θετική τροπή σε όλο αυτό το προβληματισμό. Καταρχήν, δεν ζήτησα κατάργηση των δηλώσεων. Πρέπει όμως τουλάχιστον να συζητήσουμε την περίπτωση αυτή. Γι' αυτό έβαλα το γιώτα, για να το συζητήσουμε. Σας ζητώ λοιπόν τουλάχιστον να ανταλλάξουμε απόψεις, να αρχίσουμε τη συζήτηση. Μπορούμε να αποφασίσουμε να διατηρηθούν ως έχουν, αλλά τουλάχιστον να έχει γίνει η συζήτηση στις πολιτικές ομάδες για να συμφωνήσουμε τι θα πούμε στον κόσμο. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι με τα εργαλεία αυτά, τις γραπτές δηλώσεις κλπ, γιατί έχω και μια άλλη έκθεση, όπου οι συνάδελφοι λένε ότι όσο περισσότερες γραπτές δηλώσεις γίνονται τόσο πιο ενδιαφέρουσα γίνεται η Ολομέλεια. Δεν συμφωνώ εγώ. Εμείς θέλουμε να καταπολεμηθεί η ιδέα που έχει ο κόσμος ότι δεν έχουμε τίποτε να πούμε. Ως Πολωνός που είχα πρωτοεκλεγεί στο Κοινοβούλιο νόμιζα ότι αυτό αυτή η εντύπωση υπάρχει μόνο στην Πολωνία επειδή είναι καινούργια χώρα, αλλά είδα ότι υπάρχει παντού, ότι δεν έχουμε καμιά δουλειά, απλώς γράφουμε δηλώσεις που δεν σημαίνουν τίποτα. Και για την αποτίμηση της δουλειάς μας, με το παράδειγμα της Πολωνίας το λέω αυτό, υπάρχουν βουλευτές που μιλάνε στην Ολομέλεια 150 φορές, κάνουν μία-δύο γραπτές δηλώσεις και το κοινό, μέσω των δημοσιογράφων κλπ, νομίζει ότι δουλεύουν με αυτά αποτελέσματα, ενώ δεν κάνουν καμία νομοθετική δουλειά, δεν γράφουν εκθέσεις κτλ. Γι' αυτό δεν είμαι και τόσο υπέρ των γραπτών δηλώσεων. Θέλω λοιπόν τουλάχιστον να συζητηθεί το θέμα για να δούμε αν ο κόσμος θεωρεί ότι είναι μεν σημαντικό αλλά δεν είναι η κυριότερη δουλειά που κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο γιατί είδαμε ότι ο κόσμος μας βλέπει σαν να είμαστε ακόμα στη δεκαετία του 70 ότι γράφουμε ψηφίσματα και δηλώσεις και η ίδια πρωτοβουλία χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, λοιπόν. Αυτή η διαστρεβλωμένη εικόνα θέλω να διορθωθεί. Όσο για αυτά που είπατε, με όλο το σεβασμό που οφείλω και για τις θέσεις των μειονοτήτων, δεν είναι πρόβλημα αυτό, δεν τίθεται, γιατί αν κάτι δεν υποστηριχθεί από τους μισούς βουλευτές δεν θα έχει κανένα βάρος. Αλλά για αυτά τα διακομματικά που είπατε, ότι δημιουργούν ένα πιο θετικό κλίμα, εκεί ίσως έχετε δίκιο. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να απλοποιηθεί τουλάχιστον η διαδικασία. Να μην υπάρχουν επικαλύψεις και να βρεθεί. Αν μπορεί κάτι να τεθεί πιο αποτελεσματικά να το κάνουμε έτσι. Αλέως δηλαδή. Τέλος, για τον μεγάλο αριθμό τους. αφού λέμε στο μέλλον ίσως και να τις καταργήσουμε θα πρέπει τουλάχιστον να συζητήσουμε το θέμα της απλοποίησης και της μείωσής τους. Να έχει μεγαλύτερη διακριτική ευχαίρεια ο πρόεδρος του κοινοβουλίου κλπ. Ίσως να αποδειχτεί ότι θα ήταν δύσκολη αυτή η αλλαγή. Να ξέρουμε αυτά. Μερικές φορές υπογράφουν οι συνάδελφοι έτσι γιατί ντρέπονται να μην υπογράψουν ή ντρέπονται να πούν δεν υπογράφω γιατί δεν συμφωνώ. Δεν το κάνουν όλοι. Λοιπόν, τουλάχιστον να απλοποιήσουμε, να αρχίσουμε τη συζήτηση όπως λέω στο γιώτα του σκεπτικού. Περιορισμένος αριθμός, μεγαλύτερη διακριτική ευχαίρεια για τον πρόεδρο και περισσότερο θάρρος να αρνείται. Δεν θέλω τη δουλειά μου να την κρίνουν με βάση ορισμένες γελίες δηλώσεις για μη ενδιαφέροντα θέματα. Αυτό. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με την έκθεση Ταρκόφσκι. Πρέπει να οριστεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Το γεγονό ότι θέλουμε να προχωρήσουμε ε, με παραπλάνησε και ξέχασα ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, η προθεσμία, για καταλεκτική προθεσμία, η διορία είναι 22 Μαρτίου στις 12 ε, για κατάθεση τροπολογιών έκθεση Ταρκόφσκι. Ε, νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να προβούμε και σε άλλη μια ανταλλαγή απόψεων με βάση τις ε, συγκεκριμένες απολογίες για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε στη συνεδρίαση της 19ης. Όπως σας είπα, η προθεσμία είναι 22 Μαρτίου. Δεν θα ψηφίσουμε, θα ξανασυζητήσουμε τις ε, τροπολογίες στις 19 και 20 Μαρτίου. Και μετά, αν θέλετε, ε, μπορούμε να ψηφίσουμε βέβαια και νωρίτερα. Ζητώ συγγνώμη κύριε Τακόφσκι που ξέχασα να το πω αυτό σχετικά με τις προθεσμίες. Πρόεδρε, καταρχήν συμφωνώ, δεν έχω μπροστά μου ε, την ατζέντα μου και δεν θυμάμαι τώρα πότε είναι οι διακοπές του Πάσχα. Θέλω μόνο να πω το εξής. Επειδή είναι πολύ σημαντικό να μην ε, χάσουμε αυτή τη συζήτηση και η συζήτηση να γίνει καλή, ε, τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έρθουν σε επαφή με τις πολιτικές τους ομάδες και με τους συναντέλφους τους. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτιμώ να έχουμε χρόνο. Καλύτερα να επιτρέψουμε ένα περισσότερο μήνα στον εαυτό μας, αλλά να είμαστε σίγουροι ότι είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε βάθος το θέμα στις ε, πολιτικές μας ομάδες για να ε, εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Γιατί δεν θα υπάρχει τότε να επανέλθουμε στο όλο θέμα. Σας είπα, δεν έχω μπροστά μου το ημερολόγιο. Ε, μακάρι να βολεύουν οι ημερομηνίες που αναφέρεται, αλλά καλύτερα κατά την άποψή μου να δουλέψουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γιατί έτσι θα δώσουμε και μεγαλύτερο βάρος στην όλη συζήτηση. Συμφωνώ απόλυτα, πράγματι, αυτή τη συζήτηση με την κάνουμε και με τις πολιτικές μας ομάδες. Και εγώ ε, είμαι σύμφωνος, δεν, βλέπω, λοιπόν, δεν βλέπω να ε, διαφωνεί κανείς. Μπορούμε, αν θέλετε, την ε, ε, κατάθεση, την προθεσμία, να την πάμε πότε να την πάμε να την αναβάλουμε λίγο. Α, μισό λεπτό, λέει ο συγγνώμη. Η γραμματεία μου προτείνει το εξή: Να ε, διατηρήσουμε την 22 Μαρτίου, Μαρτίου, ως καταληκτική ημερομηνία για τις προθεσμίες. Η συζήτηση να γίνει στις 26 Απριλίου και να ψηφίσουμε το Μάιο. αν μεταθέσουμε την πληροφορία, μπορούμε να μεταθέσουμε και τις ε, τροπολογίες. Κοιτάξτε, ζήτησανε ε, αρκετά ε, πλούσια αλλά έτσι γενικής φύσεως. Ίσως λοιπόν πρέπει να εκφραστούμε πιο συγκεκριμένα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω την 22 Μαρτίου για τις τροπολογίες, όπως σας είπα η τον Απρίλιο και μετά η ψηφορία τον Μάιο. Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ίσως η συνάδελφος η κυρία Γκουρμάη, ε, η αντιπρόεδρός μας, ε, μπορεί να μας ενημερώσει για τη δική της την έκθεση το σημείο υπαριθμών 9 που αφορά στην τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών. Δηλαδή, αν έχουν συγκεντρωθεί οι απαραίτητες υπογραφές, τι γίνεται μετά. τόσο, η κυρία Γκουρμάη έχει το λόγο. Καταρχά, χαίρομαι πολύ που λαμβάνω το λόγο σήμερα γιατί είναι πολλοί συνάδελφοι παρόντε και το θέμα είναι πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη γιατί στις 26 ε, Ιανουαρίου δεν ήμουν παρούσα όταν συζητήθηκε ε, η δημόσια ακρόαση και η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών και ήταν και λίγοι βουλευτές ε, παρόντες ούτως ή άλλως. Σε ό,τι αφορά πάντως τις συζητήσεις, ενημερώθηκα μετά Είχα επαφή με εκπροσώπους Επιτροπής ε, Αναφορών και άλλους βουλευτές που επίσης ε, συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή μέχρι στιγμής και κυρίως τον Γκέρχαρτ Χέφνερ. Η Νταϊάν Βόλη, όπως ξέρετε, δεν είναι μαζί μας πια. Έχουμε όμω τον Έντουαρτ Μακμίλαν Σκότ, ο οποίο επεξεργάζεται το θέμα σε συνεργασία μαζί μα. Ε, ήταν παρόν και η πρόεδρο τη Επιτροπή Αναφορών ήταν παρούσα και αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερω. Έχω μελετήσει τι διαθέσιμε πληροφορίε και έτσι μπορώ να σα παρουσιάσω σήμερα αυτό το σχέδιο. Βέβαια, και ο Αλέν Λαμασούρ ε, Σκιώδη συμφωνεί, αν και δεν είναι σήμερα εδώ, διότι έχει συναντήσει με την Εθνική Αντιπροσωπή και κάποιου Ούγγρου συναδέλφου αυτή τη στιγμή. Μια νέα εξέλιξη, την οποία ενδεχομένω γνωρίζετε, είναι ότι έχουμε πλέον αντιπρόεδρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρμόδιο για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών και συγκεκριμένα τον κύριο Παπαστάμκο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε να τον συναντήσουμε και να τον ενημερώσουμε για την όλη διαδικασία για τι ε, Πρωτοβουλίε Ευρωπαίων Πολιτών και διαισθάνομαι ότι γενικά συμφωνούν όλοι ότι θα έπρεπε να οριστεί μία μόνο θήρη, ένα one-stop shop που θα εξεργάζεται αυτές τις ε, πρωτοβουλίε, θα ανταλλάσσει απόψεις, θα ξεκινά διάλογο με τους εκπροσώπους ε, των πολιτών, των ενώσεων και βέβαια και με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ θα έλεγα. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και απαραίτητη διοικητική στήριξη και ο αντιπρόεδρος Παπαστάμκος είναι έτοιμος και διατεθειμένος να αναλάβει το ρόλο αυτό. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι θα έχουμε υψηλή εκπροσώπηση σε ό,τι αφορά τις ε, πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών, θα προεδρεύει και τις αντιπροσωπείας που θα διαπραγματεύεται με την Κομισιόν. Και έτσι υπάρχει συνεργασία με τα δύο θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά δημόσιες ακροάσεις για ECI, Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών. Συντονίζεται λοιπόν έτσι η συζήτηση και η ακρόαση και συμμετέχουν οι αρμόδιες επιτροπές. Αν χρειαστεί τώρα να υπάρξει επαφή με την Κομισιόν ή άλλα θεσμικά όργανα φορείς, θα το πράξουμε, ώστε να οργανώνονται και να διεξάγονται με το σωστό τρόπο οι ακροάσεις. Και έπειτα η αρμόδια επιτροπή είναι αυτή η οποία θα αναλαμβάνει ο διοργανώσει τη δημόσια ακρόαση στο Κοινοβούλιο. Δεδομένη βέβαια τη εμπειρία που ε, έχει η Επιτροπή Αναφορών, είναι φυσιολογικό οι συντονιστές και το Προεδρείο της Επιτροπής να συμμετέχει στη διοργάνωση των ακροάσεων. Έχουμε εδώ και μία εβδομάδα διαθέσιμη την έκθεση, το σχέδιο έκθεση. Δεν ξέρω τι διαβάσατε, τη μελετήσατε, είχατε χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω εκ των προτέρων όλους όσους θα έρθουν σε επαφή μαζί μου και αυτούς που έχουν ήδη έρθει σε επαφή μαζί μου. Σε ευχαριστώ. Αλλά μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω. Βέβαια η Ζήτα τα είπε αυτή, τέλος πάντων. Ένα σημείο θέλω κι εγώ να τονίσω. Υπήρξε μια πρόταση να υπάρχει μεγαλύτερη σάφή και τα λοιπά, να είναι μια επιτροπή δηλαδή αρμόδια, αλλά είχαμε και πιστικά επιχείρηματα από την Επιτροπή Αναφορών. Αν θέλουμε όμως να ληφθεί σοβαρή υπόψη μια πρωτοβουλία, γιατί υπάρχουν πρωτοβουλίε για διάφορα θέματα και όπως είπε και ζήτα και θέλω και εγώ να το τονίσω αυτό για να το επιβεβαιώσω, η αρμόδια, εκάστοτε αρμόδια επιτροπή είναι αυτή η οποία θα πρέπει να υποπτεύει την όλη διαδικασία. Γιατί μπορεί η πρωτοβουλία συγκεκριμένα αφορά ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε και τον αρμόδιο αντιπρόεδρο και ο πρόεδρο τη Ένωση των Πρόεδρων των ευλαμβάνεται. Άρα μπορούμε να τι εξετάσουμε τι πρωτοβουλίε σε βάθο. Αν θέλουμε λοιπόν να ασχοληθούμε σοβαρά με τι πρωτοβουλίε αυτέ των πολιτών, θα πρέπει να γίνονται συζητήσει σε μεγαλύτερο βάθο. Αυτό μπορεί να σημαίνει και μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει κοινή γνώμη, ότι μπορεί να χρειάζεται να ασχολούνται πάνω από μία επιτροπέ. Πάντω πρέπει να δώσουμε το, την εικόνα στην κοινή γνώμη, ασχολούμαστε σοβαρά με αυτές τις πρωτοβουλίες. λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν να και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Κουρμάη για όλα όσα μας πρόσφερε. Το θέμα είναι τεράστιο και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρωτοβουλία των πολιτών. Η συλλογή υπογραφών από πολλούς πολίτες πολλών χωρών για να ζητήσουν ακρόαση στο Κοινοβούλιο είναι ο τελικός σκοπός και πρέπει να το σχεδιάσουμε όπως πρέπει για να μπορέσει να στηριχθεί, να γίνει βιώσιμο αυτό το εγχείρημα. Εδώ πρόκειται για την οικοδόμηση ολόκληρου γοτφικού, ολόκληρης γοτφικής Μητρόπολης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε όλο το χρόνο που χρειαζόμαστε και να το σκεφτούμε δεόντως. Την περασμένη άνοιξη είχα κάνει ένα κατάλογο όλων των θεμάτων που τίθενται για την οργάνωση ακροάσεων. Μία έκθεση λοιπόν πρωτοβουλία, η οποία θα μα έδινε τη δυνατότητα ε, τα διάφορα θέματα να συζητηθούν σε διάφορα επίπεδα. Εγώ αυτό το έκανα το ε, φθινόπωρο γραπτά. Δυστυχώ όμω ε, δεν εγκρίθηκε και στην Επιτροπή επικράτησε η άποψη ότι θα πρέπει όλα να γίνουν με τη μορφή τροπολογίας ε, του κανονισμού. Πρέπει να σας πω, ε, ανησυχώ τώρα λιγάκι, με αυτήν την ε, πρόταση ενδέχεται να καταλήξουμε σε μια πολύ περίπλοκη ρύθμιση στον κανονισμό, ένα, μια πολύ περίπλοκη διάταξη και οι πολίτες ε, δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα. Ε, ήδη εγώ, όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών, έχω κάνει την εμπειρία ότι ακόμα και πρωτοβουλίες ε, τις οποίες επεξεργάζονται νομικοί δεν είναι κατανοητές. Εγώ λοιπόν θα προτιμούσα να συμφωνήσουμε σε σαφείς κανόνες, παραδείγματος χάρη ποια επιτροπή είναι αρμόδια, πώς ε, εκτιλήσεται η διαδικασία. Και πάρα πολλά που αναφέρονται, παραδείγματο χάρη για την ε, επιστροφή δαπανών, για, την, για ε, τον τον ορισμό της ημερομηνία για τις σχέσεις με τις επιτροπές, αυτά δεν θα ήθελα να τα ρυθμίσω με τη μορφή rules of procedure, αλλά με κάποιον άλλο τρόπο. Αυτή είναι έτσι μια γενική τοποθέτηση και το βασικό ερώτημα για το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε είναι ποιο ποια επιτροπή ή ποιο όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλείται να οργανώνει αυτές τις ακροάσεις. Και εδώ έχουμε δύο προτάσεις. Η μία είναι η πρόταση της Επιτροπής Αναφορών, δηλαδή επειδή η Επιτροπή Αναφορών είναι εκείνη η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα ασχολείται με τις αναφορές των ε, πολιτών, να αναλάβει αυτή την διοργάνωση των ακροάσεων. Και η δεύτερη πρόταση, λέει, είναι ε, η ακρόαση να διοργανώνεται από την αρμόδια επιτουσίας επιτροπή. Και τα δύο ε, έχουν επιχειρήματα που τα στηρίζουν και οι δύο προτάσεις. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πρωτοβουλία πολιτών η οποία θα τοποθετείται σε συγκεκριμένα θέματα και αυτή τι ε, θα πρέπει να συζητιέται και να απευθύνεται σε εκείνους που είναι αρμόδιοι. Πιστεύω βέβαια παράλληλα ότι αν κάθε φορά έχουμε διαφορετική επιτροπή που οργανώνει αυτές τις ακροάσεις, κάθε φορά οι πολίτες θα έχουν να κάνουν μια διαφορετική επιτροπή, αυτό δεν είναι καλό. Πράγματι η Επιτροπή ε, Αναφορών είναι εκείνη που ακούει, ε, ασχολείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τις αναφορές των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν ε, ίσως να πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση που ε, θα λέει οργανώνει η Επιτροπή των Αναφορών η Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια επί της ουσίας ή επί του περιεχομένου. Δεν ξέρω τώρα ε, πόσο λεπτομέρως θα συζητήσουμε το θέμα, αλλά πρέπει, ε, παρότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, να συνεχίσουμε αύριο τη συζήτηση. Γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ε, εδώ έχει περάσει γεννός ένας, χρόνο, ένας χρόνος περίπου. Και τώρα, για πρώτη φορά, έχουμε ε, μία αναθεωρημένη πρόταση. Η όλη διαδικασία ξεκινάει από την 1η Απριλίου και υπάρχουν πολλά που πρέπει να αισθητούν σε βάθος. Συγκεκριμένα Όργανα του Κοινοβουλίου θα αναλάβουν να συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια διοργανική συμφωνία. Θα περάσει δηλαδή μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να καταλήξουμε σε αξιόπιστες ε, ρυθμίσεις. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Και επιτρέψτε με εγώ να δείξω κάποια ερωτήματα. Παραδείγματο χάρη, κατά πόσον το 197α είναι το σωστό για τον κανονισμό. Το 42 νομίζω είναι καλύτερο. Εκεί πρόκειται για ε, διαδικασίες ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πρόκειται και για το δικαίωμα πρωτοβουλίας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την πρωτοβουλία των πολιτών έχουμε πλέον μια νέα διαδικασία το άρθρο 197α ασχολείται με ρυθμίσεις μέσα στις ίδιες τις επιτροπές και γι' αυτό, κατά την άποψή μου, δεν ενδείκνεται ιδιαίτερα. Το δεύτερο είναι το εξής. Στην πράξη, η ιδέα του αντιπροέδρου ε, που θα είναι αρμόδιος για τις ε, πρωτοβουλίες των πολιτών, αυτή την πρόταση την βρίσκω λογική. Πιστεύω όμως ότι εδώ πρέπει να ανατίθενται ή ανατίθενται στους αντιπροέδρους αρμοδιότητες που κατ' ουσίαν είναι των προέδρων. Πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε αυτό, ε, να μην καταλήξουμε σε μία ε, συμφωνία η οποία ε, θα είναι σε αντίθεση με το άρθρο 27, το 88 και το καθεξής. Έχω και πάρα πολλά άλλα να πω. Βλέπω όμως το ρολόι και δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω τι είχατε προτείνει, τι θέλετε, πώς θέλετε να συνεχίσουμε. Είχαμε πει μέχρι τις 5 να συζητήσουμε. Εγώ δεν θέλω να μονοπολώ το χρόνο. Θέλω όμως να πω ότι για μένα χρειαζόμαστε χρόνο για συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν τελειώνω αν μου επιτρέπετε, σε αυτό το σημείο ε, θέλω να ακούσω τους ε, συναδέλφους, αλλά θεωρώντας ότι πρέπει καταρχήν να συμφωνήσουμε για το πώς ε, θα συνεχιστεί περαιτέρω εξέταση του θέματος. Τι θα γίνει με τις τροπολογίες και τι θα γίνει με την πρόταση της Επιτροπής Αναφορών. Υπήρξε αυτή η συζήτηση ε, με τους εισηγητές και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών. Νομίζω λοιπόν, δεν ξέρω τώρα πώς να το διατυπώσω αυτό, αλλά θα έλεγα ότι τελικά καταβάλλονται ε, προσπάθειες να καταλήξουμε σε μία απλή ρύθμιση και αυτό θα ήταν σκόπιμο. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέλω να κάνω έκκληση να προσπαθήσουμε σε αυτή τη συζήτηση να καταλήξουμε σε συνένεση. Αυτό είναι απαραίτητο. Εγώ ίδιος έκανα μία πρόταση για το πώς μπορεί να ρυθμιστεί το όλο θέμα. Και ε, θα μου επιτρέψετε να σας στείλω αυτή την πρόταση σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ε, μέχρι τώρα το, την έστειλα μόνο στους άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά νομίζω ότι ε, τώρα μπορώ να στείλω την πρόταση αυτή σε όλους και στόχος μου είναι να καταλήξουμε σε έναν κανονισμό ο οποίος δεν θα βρίσκεται σε αντίφαση με άλλους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έτσι να αντιμετωπιστεί το θέμα. Πράγματι δεν έχουμε πολύ χρόνο, λέει ο Πρόεδρος, αλλά το όλο θέμα είναι τόσο σημαντικό, έτσι ίσως ε, θα πρέπει να το αφιερώσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μία παρέμβαση. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε σύγκριση ανάμεσα στις αναφορές και στην πρωτοβουλία των πολιτών. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και διαφορετικά τα αντιμετωπίζει η συνθήκη της Λισαβόνης. Ε, για τις ε, πρωτοβουλίες των πολιτών υπάρχουν κάποιες ε, εγγυήσει, όχι μόνο ο, ο μεγάλος αριθμός των πολιτών. Βέβαια και στις αναφορές μπορεί να υπάρχει μεγάλος αριθμό των πολιτών. Αλλά σας λέω, είναι διαφορετικά πράγματα, είναι διαφορετικά πράγματα και κυρίως διαφορετικά διότι όταν έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές, αυτό δεν υπάρχει για τις αναφορές, είναι απαραίτητο και προβλέπεται να υπάρχει ο σωστός διάλογος με τις, ε, ο δέον διάλογος αν θέλετε, με τα ευρωπαϊκά όργανα και το ανώτατο κοινοτικό ενωσιακό όργανο το οποίο ασχολείται με τις πρωτοβουλίες των πολιτών είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί το άρθρο 11 της συνθήκης λέει ότι οι πρωτοβουλίες των πολιτών αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετική πράξη. Άρα δηλαδή Ό,τι και να αποφασίσουμε ε, από τη στιγμή που έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε να συμπεριλάβουμε και να εμπλέξουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα δηλαδή το θέμα είναι ε, με ποιον θα κάνουμε το διάλογο. Εντάξει, καλό είναι το Κοινοβούλιο να τοποθετείται, αλλά το βασικό είναι ε, ποιος είναι καταρχήν αρμόδιος και αρμόδια είναι η Επιτροπή και γι' αυτό η Επιτροπή πρέπει να συμπεριληφθεί όχι τυχαία, αλλά όπως σας είπα ε, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Αυτό λοιπόν ε, που έχει σημασία είναι όπως σας είπα ότι αρμόδια είναι η Εκτελεστική Επιτροπή. Βέβαια δεν θα απέκλεια ότι προαιρετικά Οποτεδήποτε πρόκειται για μια σημαντική ε, πρωτοβουλία πολιτών, σε αυτές τις περιπτώσεις να ακολουθεί μια ε, σοβαρή συζήτηση και κατεξαίρεση στο Κοινοβούλιο. Στην Ολομέλεια μάλιστα το Κοινοβουλίου. Ναι. Αλλά εντάξει θα το σκεφτούμε αυτό. Θέλω να ξέρω να μάθω και κάτι άλλο. Αυτές ε, οι νέες εφαρμογές ε, με τις οποίες ασχολείται η κυρία Γκουρμάη ε, αφορούν το χρονικό διάστημα μετά τον Απρίλη και ένα χρόνο μετά την ε, θέση εφαρμογή όλου αυτού του σχεδίου. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό αυτή η Επιτροπή να είναι ικανοποιητικά ενημερωμένη για το τι θα συμβεί από τον Απρίλιο και μετά. Δηλαδή τους κανόνες που θα έχουν θεσπίσει οι, ε, τα διάφορα κράτη για να ε, ρυθμίζουν ε, τη συγκέντρωση των υπογραφών και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. Ίσως μπορούμε και να συζητήσουμε για το θέμα αυτό και με μία άλλη επιτροπή. Τώρα έχει ζητήσει το λόγο να μιλήσει ο κύριος Νταφ, μάλιστα. Ευχαριστώ. Πρέπει να φύγω πάρα πολύ σύντομα όμως να πω κάτι γιατί πρέπει να προχωρήσουμε κατά την άποψή μου. Έχουμε και τη συνεδρία των συντονιστών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να σεβαστεί τις δικές του αρμοδιότητες, τις νομοθετικές. Φοβούμε, μην εμπλακούμε σε πάρα πολλές ακροάσεις, σε προνομοθετική φάση, σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες των πολιτών, μήπως τελικά περιορίσουμε τη δική μας δυνατότητα ελιγμών σε κάποια μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και συμφωνώ με εσάς κύριε Πρόεδρε. Ότι η Κομισιόν έχει ευθύνη ύψιστη σε αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει να διατηρηθεί η ανεξαρτησία δράσης της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την ε, παραλαβή πρωτοβουλίων των Ευρωπαίων Πολιτών. Τέλος, Δεν μου αρέσει πολύ αυτή η διατύπωση που λέει ότι θα υπάρχει ένας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα είναι αρμόδιος για τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Γιατί οι πρόεδροι του Κοινοβουλίου είναι υπεύθυνοι απέναντι του Προεδρίου. Σε αυτό λογοδοτούν. Οι ευθύνες τους είναι ευθύνες, είναι αρμοδιότητες που τους ε, αναθέτει ή μπορεί να τους αναθέσει το Προεδρείο για κάποιους τομείς εργασίας. Δεν μπορούν να πάρουν ε, εκτελεστική αρμοδιότητα ή ευθύνη για οτιδήποτε έτσι αυτό αυτοδικαίωση. Επομένω, καλό θα ήταν κατά την άποψή μου να προσαρμόσουμε τη διατύπωση σε ό,τι αφορά την ε, θέση και το ρόλο του Αντιπροέδρου. Έχω να κάνω και άλλες παρατηρήσεις, αλλά θα το κάνω αυτό σε κάποια άλλη συζήτηση. Αλλά και εγώ συμφωνώ πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν ε, σύντομοι. Επιτρέψτε μου να πω κάτι πάρα πολύ σύντομα, γιατί αφορά στην ε, ε, διεξαγωγή των περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Είπατε ότι δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι την 1η Απριλίου, έχετε απόλυτα δίκιο και είπατε ότι αρκεί ε, να είμαστε έτοιμοι μετά από ένα χρόνο. Αυτό όμως ε, δεν ισχύει κατά την άποψή μου. Οι 12 μήνες είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα και είναι δυνατόν μετά από 2-3 μήνες ε, να έχουμε μπροστά μας μια έτοιμη πρωτοβουλία. Άρα δηλαδή πρέπει να επιταχύνουμε και όλα τα άλλα θα τα πούμε εν το χρόνο. Εντάξει κυρία Γκουρμά, εσείς έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Υπήρχε λόγος λοιπόν που ήθελα να συζητήσουμε σήμερα αυτό το θέμα επειδή είσαστε τόσοι πολλοί παρόντε, τη, Δευτέρα, τη τελευταία φορά ήταν δύο συνάδελφοι μόνο. Ούτε κι εγώ ήμουνα παρούσα και ζήτησα συγγνώμη γι' αυτό. Χαίρομαι που είσαστε εδώ λοιπόν σήμερα τόσοι πολύ και κάνετε και τα σχόλια αυτά που κάνετε. Συμφωνώ με τον Γκέρχαρτ ότι θα πρέπει να είμαστε, ε, να βιαστούμε Γι' αυτό και θα πρέπει και η προθεσμία για τις τροπολογίες να είναι 20 Μαρτίου, όπως ζητήθηκε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους, γιατί ενισχύουν τη δική μου προσέγγιση. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συμπεριλάβω όλες αυτές τις ιδέες για να είμαστε ξεκάθαροι αυτό που είπατε για τον αντιπρόεδρο θα το λάβω υπόψη μου. Πρέπει να σα πω βέβαια ειλικρινά ότι με ε, ξέπλαξε το ότι ο Μάρτιν Σούλτ ήταν αυτό ο οποίο όρισε αντιπρόεδρο υπεύθυνο για την ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών. Έδειξε αυτό ότι θεωρεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Αν ε, αναθέτει αυτό το χαρτοφυλάκιο κατά κάποιο τρόπο σε έναν αντιπρόεδρο, έτσι πρέπει να το εκλάβουμε. Το έχουμε ήδη συζητήσει, είπατε και ορισμένοι από εσάς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσκαλούνται και άλλες επιτροπές να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία της ε, πρωτοπλίας πολιτών. Αυτό άλλωστε είναι η δημοκρατία, συνάδελφοι σε διάφορες επιτροπές να μπορούν να έρχονται σε επαφή με τις ιδέες, αν θέλετε, των Ευρωπαίων πολιτών το να είναι αυτό το θέμα δεν στη διάταξη τη διάσκεψη των των επιτροπών δεν με ενοχλεί, γιατί πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη του πολίτε και τι πρωτοβουλίε του. Γιατί αν μιλάμε για ένα εκατομμύριο υπογραφέ, ε, δεν είναι κάτι αστείο και πρέπει να του δώσουμε τη δέουσα προσοχή και σημασία. Πρέπει λοιπόν να συμμετέχουν και άλλες επιτροπές γιατί ξέρουμε ότι τα θέματα μπορεί να ποικίλουν. τι έγινε στη διάρκεια αυτού του χρόνου σε σχέση με την πρώτη δημοσίευση για τι πρωτοβουλίε πολιτών. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ πρωτοβουλίες πολιτών αφενός και αναφοράς αφετέρου. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε αυτά τα δύο πράγματα να είναι ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Θα μπορούσαν οι υπογραφέ, αν δεν φτάσουν τον εκατομμύριο, μάλλον οι πρωτοβουλίε που δεν θα συγκεντρώσουν ένα εκατομμύριο υπογραφέ, να αντιμετωπίζονται ω αναφορέ. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να συνεργαστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή Αναφορών. Είναι πάρα πολύ σημαντική η Επιτροπή Αναφορών, ούτω ή άλλω. Να σας πω ότι περιμένω εξαιρετικές τροπολογίες από εσάς. Πάντοτε είμαι διτεθειμένη να εξεύρουμε καλό συμβιβασμό. Σας ευχαριστώ ήδη για τη συνεργασία. Λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα. Αν θέλουμε να ε, αντιδράσουμε με ταχύτητα, πρέπει να βιαστούμε. Άρα 6 Μαρτίου για την κατάθεση τροπολογιών, μέχρι τις 12 για να μπορούμε να ψηφίσουμε ε, στις συνεδρία τη 20 Μαρτίου. Και πρέπει να σου πω ειλικρινά ότι νομίζω είναι λίγος ο χρόνος, είναι περιορισμένος. Εάν λοιπόν ε, ε, θέλουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο, η τροπολογία στις 20, μέχρι τις 20 Μαρτίου και η ψηφορία στις 26 Απριλίου. Νομίζω ότι το δεύτερο είναι καλύτερο. Τι λέτε εσείς κυρία Γκουρμάη. Η δημοκρατία είναι αυτή η οποία πρέπει να επισχύσει, άρα πρέπει να αποφασίσουμε εδώ. Αν ο Γκέρχαρτ πιστεύει ότι πρέπει πριν την 1η Απριλίου να είμαστε έτοιμοι, τότε ναι. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αν όμω θέλετε να κάνετε και άλλα σχόλια και εξαιρετικέ τροπολογίε να καταθέσετε, α επιλέξουμε τη δεύτερη προθεσμία. Όποια εσεί κρίνετε ότι είναι η καλύτερη επιλογή για όλου. Αν θέλω να δείξω στου πολίτε μα ότι είμαστε έτοιμοι πριν την 1η Απριλίου, επιλέγουμε την πρώτη. Ε, προθεσμία. Αν όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να δεχθώ τη δεύτερη προθεσμία. Έφνερ. Ο κύριος Έφνερ, πριν ε, γίνουν ερμηνείε του τι επιθυμώ, καλύτερα να τα πω μόνο μου. Εγώ είμαι υπέρ τη ε, δεύτερη εναλλακτική λύση που μα δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε αυτό το τόσο σημαντικά. Και κατά τα άλλα, αυτά που θέλω να πω τα λέω μόνο μου. Και το λέω επειδή μερικοί ερμήνευσαν ε, ότι ε, είμαι και μέλος Επιτροπής Αναφορών και συντονιστής. Κοιτάξτε, αφήστε να τα λέω μόνος μου. Εγώ αυτά που θέλω να πω τα λέω. Ε, νομίζω ότι αυτό όλοι θα πρέπει να το κάνουμε. Η δική μου λοιπόν η προτίμηση είναι, όπως σας είπα, να έχω σήμα. Αυτό σας είπα, αν θέλετε να ασχοληθούμε για μεγαλύτερο χρόνο, κανένα πρόβλημα να μην βιαστούμε. Άρα ας κρατήσουμε τη δεύτερη προθεσμία λοιπόν. Κατόπιν τούτου, μετά από αυτά που είπε η κυρία Γκουρμάη και αυτά που είπε ο κύριος Χέφνερ, θα έλεγα ότι μπορούμε 22 Μαρτίου μέχρι τις 12 να ορίσουμε την ημερομηνία για την κατάσταση τροπολογιών και στις 26 Απριλίου ψηφίζουμε. Αυτά ε, αποφασίσαμε και έκλεισε η συνεδρίαση και έτσι μετά από ένα μικρό διάλειμμα θα πάμε στη συνεδρίαση των συντονιστών για αύριο. Θα μείνουμε να συζητήσουμε ε, την έκθεση του κυρίου Χέφνερ Ευρωπαϊκότητας των Πολιτών, έκθεση Ραντζέλ, η 5. Μετά η 6, δύο εκθέσεις έχει ο κύριος Ραντζέλ και μετά οι ψηφοφορίες. Τρεις εκθέσεις και οι ψηφοφορίες. Δέκα και μισή θα ψηφίσουμε. Εντάξει.